Ήθελα απλώς να πω ότι το Προεδρείο απουσιάζει. Γι' αυτό και μου ζήτησαν, επειδή είμαι ο πιο ηλικιωμένος, να αναλάβω προσωρινά αυτή τη θέση. Με μεγάλη χαρά βεβαίως αναλαμβάνω αυτή την αποστολή και ελπίζω να με βοηθήσετε όλοι. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης η οποία σας έχει δοθεί. Έτσι, μήπως κάποιος θα ήθελε να προβάλλει κάποια αντίρρηση. Όχι, κανείς. Υιοθετείτε λοιπόν, εγκρίνεται η διάταξη. Και τώρα τα πρακτικά της 8ης Φεβρουαρίου. 2010. Έτσι. Και στο σημείο αυτό, μήπως κάποιος θα ήθελε να κάνει κάποια παρατήρηση, ή κάτι να πει. Εγκρίνονται τα πρακτικά. Και τώρα ξεκινάμε με το επόμενο σημείο, τέταρτο σημείο. είναι η επιβολή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην εσωτερική αγορά πνευματικής ιδιοκτησίας λοιπόν και πριν να δώσουμε το λόγο στην εισηγητριά μας θα ήθελα στο σημείο αυτό να σας υπενθυμίσω ότι είναι πολύ σημαντική η σημερινή συνεδρίασή μας. Γιατί? Στις 10 η ώρα θα έχουμε μια συνάντηση για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Όπως έχει ήδη λοιπόν αναγγελθεί, πρόκειται για μια σημαντική και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία της Επιτροπής μας. Ίσως, στο σημείο αυτό, επειδή δυστυχώς έχω και σε μια άλλη συνεδρία, σε λίγο πριν 10 θα πρέπει να αποχωρήσω από την αίθουσα έτσι μη σας εκπλήξει αν δείτε κάποιον άλλο να προεδρεύει τη συνάντησή μας. Είμαι σκιώδης συγητής σε κάποια άλλη συνεδρίαση. Έχουμε δύο αντιπροέδρους που φτάνουν σε λίγο από το αεροδρόμιο. Ελπίζω να φτάσουν αρκετά νωρίς για να με αντικαταστήσουν. και θα παραδώσω τη σκητάλη στον αντικαταστάτη μου και μετά θα επανέλθω, έτσι. Το λόγο έχει η Σουζάννα Ροϊτόβα, η οποία θα μας ε, παρουσιάσει Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ καταρχήν που αναλάβατε την ε, Προεδρία αυτής της Επιτροπής, γιατί έτσι μπορούμε να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Είναι μεγάλη χαρά για μένα που μπόρεσα να προετοιμάσω αυτήν την ε, εργασία. Με ενδιαφέρει το θέμα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Καταρχήν η συνεργασία με την κυρία Γκαλό ήταν εξαιρετική από την νομική επιτροπή. Υπάρχουν ε, χιλιάδες ε, απομιμήσεις προϊόντα τα οποία μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό και θα πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, να υιοθετήσουμε πιο αποτελεσματικά εργαλεία για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Φυσικά η γνωμοδότησή μου είναι περιορισμένη και προτείνω οκτώ διαφορετικά σημεία, οκτώ σημεία τα οποία υποβάλλονται σαν συστάσεις και βεβαίως υπάρχουν και κάποιες τροπολογίες. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί η, Επιτροπή θέλει να δημιουργήσει ένα κέντρο για τις απομιμήσεις και τα πλαστά προϊόντα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, να δημιουργηθεί ένα είδος παρατηρητήριο, ένα κέντρο από το οποίο να ξεκινάει η αποτελεσματική μας δράση. Όλες αυτές οι δραστηριότητες και η δημιουργία ενός τέτοιου κέντρου θα είναι πάρα πολύ σημαντικές και θα μπορέσουν να λειτουργήσουν με αποτελεσματικό τρόπο εάν βεβαίως βασιστούμε σε ένα σχέδιο εργασίας και σε καλό συντονισμό. Το παρατηρητήριο αυτό, αυτή τη στιγμή παραδείγματος χάρη, δεν έχει επαρκή χρηματοδότηση. Απαραίτητο είναι ο αρμόδιος για το κέντρο αυτό, δηλαδή η Επιτροπή να αναλάβει το θέμα της χρηματοδότησης. Το κέντρο αυτό θα εργάζεται όχι μόνο στα προϊόντα τα οποία είναι απομιμήσεις, τα οποία δεν είναι γνήσια, αλλά και για κάθε άλλου είδους τέτοιες ε, διαδικασίες πλαστογραφίας, απομίμησης. διπλώματα έβρεση τεχνίας, μάρκες, προστασία σημάτων στο πνευματικό και στον υλικό τομέα. Δικαιώματα δηλαδή διανοητικά, διανοητικής ιδιοκτησίας στην εσωτερική αγορά. Θα πρέπει επίσης να επικεντρωθούμε και σε ψηφιακά προϊόντα. Είναι εκατομμύρια τα προϊόντα, τα πλαστά, τα μιγνήσια τα οποία μπαίνουν από τρίτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε με αυστηρό και αποτελεσματικό τρόπο το φαινόμενο αυτό. Ζητώ λοιπόν από την Επιτροπή να συνεχίζετε τις προσπάθειές της έτσι ώστε αυτό το παρατηρητήριο να γίνει αποτελεσματικό και να μπορέσει να έχει άμεσα αποτελέσματα. Κάνω μια έκκληση εδώ προς την Επιτροπή, η οποία ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία, έτσι ώστε να αναθεωρηθεί η παρούσα νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ένα μεγάλο αριθμό μη γνήσιων προϊόντων που μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν πραγματικά να δούμε πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά, τους νέους καταναλωτές, όσον αφορά αυτά τα προϊόντα απομίμησης. Υπάρχουν πολλές φορές παραδείγματος χάρη και επικίνδυνα προϊόντα, επικίνδυνα για την υγεία. Γι' αυτό και για τα παιχνίδια παραδείγματος χάρη οι κανόνες πρέπει να γίνουν πάρα πολύ αυστηροί. Το ίδιο και για τα φάρμακα, το ίδιο και για τα είδη διατροφής. Τρεις τομεί που έχουν άμεση επίπτωση ε, στην υγεία. Για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας η Επιτροπή θα πρέπει να περάσει αμέσως, το 2010 δηλαδή, στις εφαρμοστικές διατάξεις, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα της υπάρχουσας νομοθεσίας. Κατόπιν στις προτάσεις μου λέω ότι αν θέλουμε να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα όλων αυτών των προσταθεών, θα πρέπει να λειτουργήσει ένα νομικό πλαίσιο με παραδείγματος χάρη πιστοποίηση πιστοποιητικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προστασία των σημάτων που σήμερα είναι κάτι που γίνεται με πάρα πολύ ελληπή τρόπο. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε και κάποια εργαλεία τα οποία υπάρχουν στους διεθνείς κανόνες που ισχύουν σήμερα για τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές. Υπάρχουν σήμερα πιστοποιητικά και προστασία των σημάτων τα οποία θα πρέπει να συμπληρωθούν από την ευρωπαϊκή, από την κοινοτική νομοθεσία. Αυτό θα πρέπει να μας επιτρέψει να προστατεύσουμε τον κόσμο των επιχειρήσεων, να δώσουμε στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, στις ευρωπαϊκές εταιρείες ένα εργαλείο τον οποίο να μπορεί να το χρησιμοποιήσει ε, στις διεθνείς τις συναλλαγές. Αυτό δεν πρόκειται να έχει απολύτως καμία οικονομική επίπτωση για τον ε, κοινοτικό προϋπολογισμό. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις και το κέντρο του Αλικάντε. Τα κράτη-μέλη λοιπόν θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη να ενδυναμωθεί αυτή η νομοθεσία, αυτές οι ρυθμίσεις θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλοι οι υπάρχοντες οργανισμοί στα κράτη-μέλη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να μην υπάρχει απολύτως καμία επικάλυψη. Προτείνω επίσης ε, μέτρα για την προστασία των καταναλωτών και στο άρθρο 18 ε, του Κανονισμού για την Προστασία των Καταναλωτών του 2004 προτείνουμε συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών οργανισμών και οργανισμών που υπάρχουν στις τρίτες χώρες με κυρώσεις όσον αφορά τις απομιμήσεις. Και βεβαίως μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και ο τομέας του ηλεκτρονικού εμπορίου, e-commerce. Στην έκτη σύστασή μου αναφέρω όλα αυτά τα προϊόντα που έρχονται από τρίτες χώρες, τα, τις απομιμήσεις που προέρχονται από τρίτες χώρες. Στο σημείο 18 και στο σημείο 10 αναφέρομαι στις διαπραγματεύσεις που ήδη έχουν ξεκινήσει μεταξύ της Επιτροπής και στις οποίες το άρθρο αυτό δεν συζητείται με ανοιχτό τρόπο αν θέλετε. Ε, υπάρχουν επίσης και οι αρνητικές απομιμήσεις αυτών των προσπαθειών ρύθμισης όπως παραδείγματο χάρη για τον τομέα των ψηφιακών προϊόντων. Οι επιπτώσεις της προστασίας, αν θέλετε, των ε, συγγραφέων, των καλλιτεχνών, των δημιουργών. Ξέρουμε ότι το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ λεπτό και θα πρέπει να συζητηθεί ακόμα περισσότερο. Η δημιουργικότητα, η προστασία της δημιουργίας, αλλά και τα όρια που θέτουμε προσπαθώντας να προστατεύσουμε αυτά τα προϊόντα, τα πνευματικά. Ξέρω ότι η γνωμοδότηση της ε, Νομικής Επιτροπής έχει επικεντρωθεί ακριβώς σε αυτό το σημείο. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε ότι υπάρχει και η εξωτερική διάσταση αυτών των προσπαθειών, κάτι το οποίο δεν έχει αντιμετωπίσει καθόλου η Επιτροπή. Το θέμα της πειρατείας. Το θέμα της πειρατείας είναι κάτι που είναι εκτός της λογικής, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων θέλει να ασχοληθεί με το κομμάτι αυτό της πειρατείας. Και τέλος θα αναφερθώ στην αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων πολλών προϊόντων τα οποία έχουν κατασχεθεί από μιμήσεις που αυτή τη στιγμή βρίσκονται κάπου σε έναν αποθηκευτικό χώρο και το κόστος είναι τεράστιο αυτή τη στιγμή. Πρέπει να μας απασχολήσει λοιπόν και η περαιτέρω χρήση αυτών των προϊόντων. Αν καταστρέφονται, πώς καταστρέφονται, αν υπάρχει περίπτωση ανακύκλωσης και τι πρέπει να γίνει. Ευχαριστώ πολύ όλους όσους με βοήθησαν τον κύριο Χάρμπερ και ευχαριστώ όλους όσους εδώ και πολλά χρόνια έχουν ασχοληθεί με το θέμα αυτό και με έχουν βοηθήσει με τις ιδέες τους. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ζητώ συγγνώμη γιατί άργησα. Θα αναλάβω την Προεδρία, προσωρινά και εγώ. Θα ήθελα να καλωσορίσω την κυρία Κωνστός Λεγκρίπ, η οποία είναι εδώ εκ μέρους του κ. Μπανία. Κυρία Ράπτη, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Όπως ευχαριστώ και τον ε, προηγούμενο Πρόεδρο, τον Αντώνιο, που μας έδωσε την ευκαιρία να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Ε, πριν ξεκινώ, ε, ξεκινήσω την παρέμβασή μου, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ρόιτοβα για την δουλειά που έχει κάνει μέχρι τώρα και να πω ότι έχω παρακολουθήσει την πορεία της και το γεγονός ότι προέρχεται και έχει εργαστεί στον ιατρικό χώρο με κάνει να πιστεύω ότι έχει αυξημένη ευαισθησία για αυτό το πολύ πολύ σημαντικό ζήτημα που αφορά τους καταναλωτές, τους πολίτες ε, δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε όσα σωστά προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως είναι ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας που υπάρχει ή η ενίσχυση της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των εθνικών διοικήσεων, παρά μόνο σε ένα σημείο προκειμένου να ενισχύσω τις προθέσεις της Επιτροπής πιστεύω ότι η επιτροπή δεν πρέπει να λειτουργεί απλώς ως ένας διαμεσολαβητής στο διάλογο μεταξύ όλων όσων έχουν όφελος από, το, από την καταπολέμηση της παραχάραξης προκειμένου να υπάρξουν αυτοδεσμευτικές συμφωνίες αλλά μάλλον να είναι η ίδια η επιτροπή που θα καλέσει που θα καλέσει τα διάφορα μέρη, ίσως μιλάω λίγο γρήγορα, ζητώ συγγνώμη, θα προσπαθήσω να μιλήσω σε αργότερο ρυθμό για να διευκολύνω και τους μεταφραστές αλλά μάλλον να είναι η ίδια η επιτροπή που θα καλέσει τα διάφορα μέρη να πάρουν μέρος στο διάλογο αυτό και στη συνέχεια βεβαίως να τον διευκολύνει. Θέλω να αναφερθώ τώρα στα σημεία του σχεδίου της γνωμοδότησης, τα οποία βρίσκω ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, αλλά και να πάρω την ευκαιρία για να ζητήσω από την εισηγήτριά μας, από την κυρία Ρόιτοβα, να μας δώσει μερικές ε, διευκρινήσεις σε κάποια άλλα σημεία. Ε, θα διατυπώσω τέλος κάποιες αρχικές πρώτες σκέψεις σε σχέση με την κατεύθυνση των τροπολογιών που προτίθεμε να κάνω. Είμαι απολύτως σύμφωνη με την πρόταση της συντάκτριας γνωμοδότησης για να ενισχυθεί η υφιστάμενη νομοθεσία. Μιλάω για την δεύτερη πρόταση και φαντάζομαι πως η κυρία Ροήτοβα εννοεί στην κατεύθυνση του να θεσπιστούν ε, ποινικοί κανόνες γιατί από τη στιγμή που μιλάμε για απώλεια ανθρώπινων ζώων ένα παράδειγμα είναι που το γνωρίζει πολύ καλά η εισηγήτρια ε, στην παραχάραξη φαρμακευτικών προϊόντων ας πούμε φοβούμε πως η απόδοση απλώς ενός προστίμου δεν επαρκεί, δεν είναι αρκετό μέτρο για να αποτρέψει ή να συμμορφώσει αυτούς που κάνουν την παράβαση βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα την πρόταση για αναλογικά μέτρα. Μιλάω για την έβδομη πρόταση. Ε, αναλογικά μέτρα για την αποτελεσματική και επιτυχή διαχείριση του αρνητικού αντικτύπου από την καταπολέμηση παραβίασης δικαιωμάτων διανοητικής ε, ιδιοκτησίας στο ψηφιακό περιβάλλον. Ε, νομίζω ότι εδώ πρέπει να δώσουμε περισσότερη προσοχή στο σχεδιασμό αυτών των μέτρων ώστε να μην δημιουργούν άλλου είδους αδικίες. Ε, θα παρακαλούσα την εισηγήτρια να μας δώσει κάποιες διευκρινήσεις σε σχέση με το σήμα πιστοποίησης της Ένωσης, την τρίτη πρόταση. Ε, σκέφτομαι, για παράδειγμα, ότι υπάρχει ήδη το περίφημο σήμα, το EC, για το οποίο έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις και το οποίο δυστυχώς κατά τη γνώμη μου δεν έχει αποδειχθεί τόσο επιτυχές όσο αρχικά φανταζόμασταν και ελπίζουμε, θέλουμε να πιστεύουμε ότι η δημιουργία ενός ακόμη σήματος ε, θα μπορέσει να βοηθήσει. Δεν θα είναι άλλο ένα ακόμη σήμα, αλλά θα μπορέσει να έχει ένα αποτέλεσμα. Πώς, ε, θα ήθελα να ξέρω τη σκέψη της εισηγήτριας πώς σκέφτεται αυτό το σήμα να λειτουργήσει αποτελεσματικά και εδώ, αν μου επιτρέπετε, να ανοίξω μία μικρή παρένθεση, επειδή έχουμε στην απογευματινή συνεδρίαση και το θέμα που χειρίζεται με πολλή επιτυχία η συγγήτριά μας, η κυρία Σαλντεμό σε σχέση με, τα, με τη σήμανση των προϊόντων. Ε, φανταστείτε ε, τα προϊόντα που πια νομίζω ότι δεν θα υπάρχει χώρος στις συσκευασίες για να μπουν τα σήματα. Ε, το λέω καθ' υπερβολήν, αλλά θέλω να δείξω ότι πραγματικά πρέπει να βάζοντας ένα σήμα να διασφαλίζουμε ότι θα έχουμε αποτέλεσμα. Ε, έχω ένα, πώς να το πω, να το πω φόβο επιφύλαξη σε σχέση με την, ε, σε σχέση με την 8η πρόταση. Μήπως ανοίξουμε ένα παράθυρο σε σχέση με τη χρήση των αγαθών αυτών. Νομίζω προς οποιοδήποτε μέτρο ληφθεί σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να σχεδιαστεί πάρα πολύ προσεκτικά ώστε να μην ενθαρρύνει με κανένα τρόπο τους παραχαράκτες να εκμεταλλευτούν τα προϊόντα αυτά αισθάνομαι την ανάγκη να κάνουμε μια μεγαλύτερη αναφορά στο κείμενο και περισσότερο έντονη σε σχέση με την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών. Με την, σε, σχέ, ναι, σε σχέση με την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών. Τους καταναλωτές έχω στο μυαλό μου ότι θα πρέπει να τους κάνουμε συμπροταγωνιστές στην καταπολέμηση της, χαρακα, της παραχάραξης. Ε, άρα οφείλουμε να τους δώσουμε μια ε, καλή πληροφόρηση, μια πολύπλευρη πληροφόρηση, συνεχή πληροφόρηση και το κυριότερο ανανεούμενη πληροφόρηση. Ε, να μπορούμε να παίρνουμε τις καινούργιες πληροφορίες και να τις δίνουμε. Αυτό το τελευταίο έχει ιδιαίτερη σημασία για τις μικρές ηλικίε. Ε, θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε μία σκέψη την οποία έχω την αίσθηση ότι πρέπει οπωσδήποτε να έχει κάνει η κυρία Ρόιτοβα ε, αν στόχος μας είναι πάντα το να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, νομίζω πως θα πρέπει να τις βοηθήσουμε σε σχέση με την εκπαίδευση και τη γνώση για τα συστήματα κατοχύρωσης δικαιωμάτων. Και για να είμαι σύντομη, τελειώνοντας, επιτρέψτε μου μία κουβέντα για την πραγματική δικαίωση των ανθρώπων εκείνων πέρα από τους καταναλωτές, για τους οποίους επίσης θεσπίζεται αυτή η νομοθεσία. Μιλάω για τους δημιουργούς. Ε, νομίζω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε όλους αυτούς τους ελέγχους που θα προχωρήσει και στις εκθέσεις που θα συντάξει, θα πρέπει να ασχοληθεί και με το θέμα της σωστής επιστροφής των ωφελών από τα δικαιώματα στους α, δημιουργούς τους. Είναι μια πρώτη σκέψη που καταθέτω εδώ ενώπιόν σας, η οποία νομίζω ότι θέλει περισσότερη έρευνα, περισσότερη δουλειά. Ε, όπως είπα και ξεκινώντας, είναι κάποιες πρώτες σκέψεις, είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα, ε, αφορά α, τους πάντες και ε, νομίζω ότι διατρέχει οριζόντια κάθε δράση η οποία συμβαίνει μέσα στην, στον επιχειρηματικό ε, χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ και πάλι την εισηγήτρια και θέλω να πω ότι είμαι στη διάθεσή της να συζητήσουμε και να βρούμε μαζί οποιασδήποτε λύσεις και βελτιωτικές προτάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you, Mrs. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Ράπτη. Δεν ξέρω ποιος άλλος θέλει να μιλήσει. Ο κύριος Κρόισμαν στη Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λίγες παρατηρήσεις ήθελα να κάνω όσον αφορά την πνευματική διανοητική ιδιοκτησία. Η παραβίαση της είναι παραβίαση ενός βασικού δικαιώματος. Πρόκειται για την παραγωγή, τη δημιουργία, από την οποία καλείται να ζήσει ο δημιουργός, ο συγγραφέας και γι' αυτό και χρειάζεται προστασία. Είναι βασικό θεμελιώδες δικαίωμα το οποίο καλούμαστε να προστατεύσουμε. Έχει δίκιο εδώ η εισηγήτρια η οποία προτείνει ένα νέο σύστημα πιστοποίησης. Το θέμα είναι, ναι, μπορούμε να συμβάλλουμε με αυτό το νέο σήμα, αυτή τη νέα πιστοποίηση. Είδαμε όμως ότι μέχρι τώρα το σήμα EU δεν κατάφερε να προστατεύσει ικανοποιητικά. Θα πρέπει λοιπόν να θέσουμε και ε, δίπλα σε αυτή τη νέα πρόταση για ε, ευρωπαϊκό σήμα και ένα σύστημα προστασίας αποτελεσματικό. Εγώ απογοητεύομαι ακούγοντας τις προτάσεις ε, της Επιτροπής και της αρμόδιας, του αρμόδιου υπότροπου. Πραγματικά θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί όταν παίρνουμε κάποιες αποφάσεις, όταν αποφασίζουμε κανόνες και ρυθμίσεις, είμαστε αρμόδιοι για την τήρησή τους. Αυτό είναι το πρόβλημα, αυτή είναι η αδυναμία μέχρι τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μη παρακολούθηση μετά την θέσπιση των κανόνων. Δεν υπάρχει παρατήρηση, δεν υπάρχει έλεγχος και εκεί είναι η αδυναμία μας. Θεωρώ λοιπόν ότι χρειάζεται ανταλλαγή πληροφοριών, στοιχείων μεταξύ όλων των φορέων και οργανισμών προστασίας των καταναλωτών και σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ την εισηγήτρια γιατί μιλήσατε για πολλά θέματα στον χώρο των ιδιών διατροφής, στα πνευματικά δικαιώματα. Όντως το θέμα αυτό περνάει όλους τους τομείς και αφορά όλους τους τομείς. Είναι λοιπόν πολύ ενδιαφέρον το ότι έχουμε αυτό το κέντρο στο Αλικάντε. Έχετε δίκιο που λέτε ότι πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε, αλλά όσον αφορά τα σήματα, παραδείγματος χάρη, ξέρετε ότι η εγγραφή στα κοινοτικά, στα ευρωπαϊκά μητρώα είναι πάρα πάρα πολύ ελλειπής. Ας στηρίξουμε λοιπόν αυτή την πρότασή σας για νέα πιστοποίηση, νέο σήμα, αλλά ακόμα πιο σημαντικό από αυτό είναι η παρακολούθηση. Παραδείγματος χάρη, πρέπει να μειωθούν πάρα πολύ τα τέλη για την εγγραφή στα κοινοτικά μητρώα. Αλλιώς θα παραμείνουν πάρα πάρα πολύ λίγα τα σήματα που θα κατοχυρώνονται. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω στην ε, εισηγήτρια ότι θα πρέπει αυτή η τελευταία μου πρόταση να συμπεριληφθεί στις ε, προτάσεις σας. Οι εθνικές αρχές, οι εθνικοί οργανισμοί θα πρέπει πραγματικά να ξεκινήσουν μια πραγματική συνεργασία με τους άλλους εθνικούς οργανισμούς. Να ξεπεραστούν τα εθνικά σύνορα, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει πραγματική ανταλλαγή πληροφοριών για το θέμα αυτό, άρα δεν μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί στην παρακολούθησή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κρόισμαν, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Έγκστρομ έχει το λόγο. με oh, Έχω διάφορα σημεία που θέλω να θίξω. Καταρχάς κάτι που συζητήσαμε πολύ στην Επιτροπή Τζούρι. Το πρόβλημα ε, της ανακοίνωσης αυτής της Επιτροπής είναι ότι μπερδεύει δύο διαφορετικά πράγματα. Από την άλλη, μία την παρατήρηση των αγαθών που όλοι θεωρούμε ότι είναι κακό και από την άλλη την παραβίαση διανοητική ιδιοκτησία στο διαδίκτυο. Αυτά είναι δύο διαφορετικά πράγματα και πρέπει να αντιμετωπίζονται ξεχωριστά. Να μην υπάρχει καμία αλληλοεπικάλυψη, ας πούμε, μεταξύ τους. Ας πούμε, η ανταλλαγή ε, αρχείων στο ίντερνετ ε, ε, και αυτός ο τρόπος πειρατεία είναι ένα αντιφατικό θέμα που πρέπει να συζητηθεί. Όταν μιλάμε τώρα για την παραποίηση προϊόντων, όλοι συμφωνούν, ακόμα και οι πειρατές, ότι πρόκειται για ένα κακό πράγμα. Αν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να ενισχύσει την πάταξη της ε, παραποίησης ε, αγωθών, ε, δεν είναι σίγουρο ότι ο καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να δημιουργηθούν νέες παράλληλες δομές. Έχουμε ήδη την Europol και έχουμε και διάφορες μορφές συνεργασίας μεταξύ των τελωνιακών αρχών των κρατών μελών. Για μένα λοιπόν θα ήταν πιο λογικό η πάταξη των παραποιημένων προϊόντων να ανατεθεί στις υφιστάμενες δομές. Είναι εύκολο για τους πολιτικούς κάθε φορά που υπάρχει ένα πρόβλημα να δημιουργούν κάτι καινούριο αντί να εξετάζουν το τι υφίσταται και να το ενισχύουν. Αυτό είναι το πρώτο θέμα που ήθελα να εγείρω, μάλλον τα δύο πρώτα θέματα. Να ε, διαχωρίσουμε αυτά τα δύο σημεία και να χρησιμοποιήσουμε τις υφιστάμενες δομές. Ένα τρίτο θέμα, στο οποίο θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας, είναι ότι υπάρχει ήδη παρατηρητήριο. Η Κομισιόν έχει ήδη ε, δημιουργήσει αυτό το παρατηρητήριο πριν καν ρωτηθεί το Κοινοβούλιο. Και αυτό ε, το θεωρώ ως ασέβεια απέναντι στο Κοινοβούλιο. Αν θέλουν τη γνώμη μας, γιατί δεν την περιμένουν τουλάχιστον και ήδη ιδρύουν το παρατηρητήριο. Αυτό με ανησυχεί. Το επόμενο θέμα για το άκτα πάλι, τη σύμβαση. Συμφωνώ με, τον, ε, με την εισηγήτρια ότι η Κομισιόν θα πρέπει άμεσα και πλήρως να ενημερώνει το Κοινοβούλιο για τις διαπραγματεύσεις. Πολύ καλό αυτό το σημείο. Ειδικότερα όσον αφορά και τη συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία δίνει στο Κοινοβούλιο αυτό το δικαίωμα. Θα ολοκληρώσω με ένα ο σημασία ε, θέμα. Δεν κατονοώ την παράγραφο 3 για αυτά τα σήματα πιστοποίησης. Ε, στην Ευρώπη ήδη έχουμε ε, μια νομοθεσία για αυτά τα σήματα πιστοποίησης. Αυτό λειτουργεί ως ένα κανονικό εμπορικό σήμα. Η καταχώρηση γίνεται με παρόμοιο τρόπο. Όμως, το σήμα πιστοποίηση σημαίνει ότι οποιοδήποτε πληρεί δεδομένα κριτήρια μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Ήδη υπάρχει αυτή η νομοθεσία. Υπάρχει ο Οργανισμός για την Εναρμόνιση της Εσωτερικής Αγοράς, είναι το γραφείο για τα εμπορικά σήματα στο Αλικάντε, εκεί μπορεί να γίνει καταχώρηση. Επιπλέον, κάθε κράτος μέλος έχει τέτοια συστήματα καταχώρησης. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν Τι θα πρέπει να προσθεθεί εδώ. Πραγματικά θα ήμουν ευγνώμων στην συγκήτρια αν μπορούσε να μας αναπτύξει λίγο περαιτέρω αυτό το θέμα. Η κυρία Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ. Θα... Αν ξεκινήσω με το τελευταίο θέμα που ανέφερε και η κυρία Ράπτη, το σημείο 3 για το σύστημα πιστοποίησης της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Θα ήθελα λίγες περισσότερες πληροφορίες από την εισηγήτρια. Τι εννοεί, υπάρχουν ήδη συστήματα πιστοποίησης. Εδώ έχουμε το πρόβλημα ότι ε, δεν γίνονται σεβαστά αυτά τα συστήματα. Υπάρχουν λοιπόν άλλες ανάγκες και δυνατότητες. Έχουμε αυτήν την υπηρεσία στο Αλικάντε και άλλες που βρίσκονται ε, εκεί. Ένα άλλο θέμα που θεωρώ ότι είναι σημαντικό και λείπει και το ανέφερε και ο κύριος Κρόιτσμαν, είναι η παρακολούθηση της αγοράς, η εποπτεία της αγοράς. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να μην είμαστε υπεύθυνοι για αυτή την εποπτεία, όμως είμαστε υπεύθυνοι ώστε να διασφαλίσουμε ότι λειτουργεί η εποπτεία. Και υπάρχουν διάφορα μέσα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Ας πούμε η συνεργασία σε τελωνιακό επίπεδο. Θα ήθελα να ακούσω τι θέλετε και εκεί να γίνει, γιατί αυτό θα ήταν μια βελτίωση που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την πειρατεία και την παραποίηση ε, προϊόντων που έρχονται έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι που λείπει λοιπόν από αυτά που μας αναφέρετε. Και ένα τελευταίο σημείο είναι ε, αφορά στο σημείο 8. Είμαι λίγο σκεπτική, όπως είπε και η κυρία Ράπτη, σχετικά με το τι εννοείται, αν θα ήταν αντιπαραγωγικό τα παραποιημένα αγαθά που έρχονται στην αφορά, αγορά ε, να διευκολύνονται με, μέσα από ε, κοινοφελείς οργανισμούς στην επαναχρησιμοποίησή τους δεν μπορείτε λίγο να μας πείτε λίγο περισσότερο τι εννοείτε με αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε την κυρία και ε, τον κύριο Σφάμπε. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εξαίρετη πρότασή της. Είναι μια βάση για μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και εγώ συμφωνώ και με ενδιαφέρει να μάθω περισσότερα γι' αυτό το σήμα πιστοποίησης και το σύστημα και το σημείο 3 που μπορεί να συμβάλλει σε αυτό ε, να υπάρχει προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας όχι μέσα στην εσωτερική αγορά μόνο αλλά και πέρα από αυτή και να ενισχυθεί και μετά υπάρχει και το θέμα του παρατηρητήριου στο σημείο 7 υπάρχει αυτή η πρόταση για τις άδειες ε, καταποκοπήν ε, πώς αυτό θα λειτουργήσει. Θα ήθελα όμως παρόλα αυτά να ευχαριστήσω την κυρία Ρόιτοβα για την πολύ καλή αυτή ε, βάση συζήτησης. Ευχαριστούμε πολύ. Επειδή δεν έχουμε πολύ ε, χρόνο και θέλουμε να τελειώσει η συζήτηση, παρακαλώ να είστε σύντομοι. Η Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Εκ μέρους της Επιτροπής να πω ότι καταρχάς χαιρόμαστε ιδιαίτερα που η Επιτροπή σας ε, μας δίνει ε, τροφή για την έκθεση της Επιτροπής ε, Τζούρι. Η Κομισιόν θεωρεί ότι δεδομένης της σημασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και του αυξημένου κύματος της παραποίησης ε, και της πειρατείας θα πρέπει το θέμα να εξεταστεί από όλες τις πλευρές ε, και να συζητείτε τακτικά στην Επιτροπή σας. Η Επιτροπή θεωρεί πως η κυρία Ρόιτοβα ε, έχει συντάξει ένα εξαίρετο σχέδιο έκθεσης και είμαστε ευγνώμονες αναφορικά με τις προτάσεις της. Η Κομισιόν ιδιαίτερα ευγνωμονεί την, υποστήρι... την κυρία Ρόιτοβα για την υποστήριξή της σχετικά με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για ε, την καταπολέμηση της ε, παραποίησης και της πειρατείας. Αυτό το παρατηρητήριο υπάρχει, αλλά είναι ένας απλός πυρήνας. Ε, χρησιμοποιείται από τη Γενική Διεύθυνση της Αγοράς για το, ως μέσο επιβολής και για να μπορέσει να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο πολιτικής είναι απαραίτητο να υπάρχουν πιο σημαντικές ανεξάρτητες και μακροπρόθεσμες δομές στο μέλλον. Αν το Κοινοβούλιο υποστηρίξει αυτή την ιδέα, η Κομισιόν είναι πρόθυμη να εξετάσει τρόπους ε, για να διασφαλίσει μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και μια ανεξάρτητη δομή για αυτό το παρατηρητήριο. Και ειδικότερο είναι κάτι το οποίο στο μέλλον θα μπορούσε να αναλάβει το Γραφείο Εμπορικών Σημάτων στο Αλικάντε. Η Κομισιόν επίσης είναι πολύ ευγνώμων για την ε, έμφαση που έδωσαν η κυρία Ρόιτοβα και η κυρία Ράπτη ε, στην ανάγκη να μάθουμε περισσότερα και να αντιμετωπίσουμε και τους ε, κινδύνους ε, για την υγεία που προέρχονται από την παραποίηση και την πειρατεία. Πρόσφατες εκτιμήσεις έχουν αποδείξει ότι το παγκόσμιο εμπόριο ε, παραποιημένων και ψευδών φαρμάκων ανέρχεται σε πάνω από 10 αμερικανικά δολάρια και αυτό δείχνει πόσο επικίνδυνη γίνεται η παραποίηση και η πειρατεία. Όχι μόνο για την ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά και για την υγεία και ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών. Η Κομισιόν επίσης ε, να καθησυχάσει το Κοινοβούλιο ότι έχει ξεκάθαρη πρόθεση στο μέλλον να ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο και να το εμπλέκει στις ε, διαπραγματεύσεις για την ε, σύμβαση, τη συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης και της απομίμησης. Υπάρχουν ανησυχίες για έλλειψη διαφάνειας σε αυτές τις διαπραγματεύσεις από την πλευρά του Κοινοβουλίου. Η Κομισιόν σας ενημερώνει ότι την επόμενη εβδομάδα στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας θα υπάρξει ένα ψήφισμα από τα κράτη-μέλη για την καταπολέμηση της παραβίασης και της απομίμησης ε, και της πειρατείας στην εσωτερική αγορά και εκεί θα τονιστεί ιδιαίτερα η ανάγκη να ε, συνεχιστεί και να γίνεται μεγαλύτερη χρήση των διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Κομισιόν επίσης ε, συμφωνεί με την κυρία Ρόιτοβα ότι πρέπει να εξετάσουμε το πώς θα ενισχύσουμε το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ε, στην φάση προετοιμασίας μίας έκθεσης ε, εφαρμογής ε, της οδηγίας εφαρμογής που θα ολοκληρωθεί μέσα στο έτος. Η Κομισιόν επίσης συμφωνεί με την κυρία Γκέπχαρτ και τον κύριο Κρόιτσμαν για την ανάγκη για καλύτερη εποπτεία της αγοράς και ένας από τους στόχους της διοικητικής συνεργασίας που προτείνει η Επιτροπή θα είναι η δημιουργία ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης μεταξύ των κρατών μελών που θα διασφαλίζει ότι όποτε υπάρχουν παραποιημένα προϊόντα στη μία αγορά, τα κράτη-μέλη, οι άλλες ε, αγορές, οι άλλες αρχές θα ε, ε, προειδοποιούνται έγκαιρα ώστε να καταστρέφονται τα προϊόντα αυτά. Τέλος, η Κομισιόν, λυπάται όμως δεν θεωρεί ότι είναι κατάλληλο να γίνει διαχωρισμός μεταξύ της παραβίασης προϊόντων και της πειρατείας ε, περιεχομένου προστατευόμενου από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Δεν έχει μεγάλη διαφορά είτε αγοράζεις ένα ε, πειρατικό CD, DVD, είτε κατεβάζεις ή ανεβάζεις ένα πειρατικό φιλμ ή ένα κομμάτι μουσικής στο ίντερνετ. Είδα κύριε Πρόεδρε το σήμα που μου κάνατε, σταματώ εδώ και ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε. Τώρα ζητώ στην κυρία Ρόιτοβα να ανακεφαλαιώσει. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να σας πω ότι επειδή ξεκινήσαμε 15 λεπτά αργότερα, περιορίστηκε και ο χρόνος συζήτησης τη εκθεσή. αυτή. Αυτό είναι πολύ ε, κρίμα. Περιοριζόμαστε επίσης και από τις ε, αρμοδιότητες της Επιτροπής μας που είναι εξορισμού ελλειπής. Γι' αυτό και πολλά από τα θέματα που θα έπρεπε να μας απασχολήσουν δεν μας απασχολούν. Είναι αρμοδιότητες της Νομικής Επιτροπής. Θα τα λέω αυτά Απλώς για να επικεντρωθώ σε τρία σημεία και να απαντήσω σε τρεις ερωτήσεις. Καταρχήν, το σημείο 7 και 8. η δυνατότητα παραδείγματος χάρη να χρησιμοποιήσουμε ένα μπλουζάκι με ένα λόγο για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν υπό κάποιες προϋποθέσεις, υπό όρους. Ότι δηλαδή αυτός ο οποίος έχει υποβάλει το σήμα, έχει κατοχυρώσει ένα σήμα, συμφωνεί. Αυτός ο οποίος κατέχει το προστατευμένο λόγο ή σήμα, επιτρέπει την χρησιμοποίηση αυτού του σήματος. Είναι δηλαδή κατά κάποιο τρόπο μία διαφήμιση που γίνεται με πλάγιο τρόπο σε κάποιον. Αυτό το λέω απλώς για να καθησυχάσω αυτούς οι οποίοι δεν θέλουν να χρησιμοποιηθούν, να ξαναχρησιμοποιηθούν, να ε, διατεθούν αυτά τα ήδη υπάρχοντα και κατασκευασμένα προϊόντα. Το θέμα τώρα του παρατηρητήριου, ένα άλλο σημείο το οποίο θα πρέπει να ε, συζητήσουμε. Υπάρχει αυτή τη στιγμή η Europol, υπάρχει η Eurojust, υπάρχουν οι τελωνιακές αρχές που συνεργάζονται, των οποίων όμως η συνεργασία θα πρέπει να ενδυναμωθεί. Βλέπουμε διαρκώς τον αριθμό των παραποιημένων προϊόντων να αυξάνεται. Χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερα μέσα, περισσότερα εργαλεία Γι' αυτό και αυτό το παρατηρητήριο θα πρέπει να γίνει με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο, με εξειδικευμένους ανθρώπους και υλικό, με σταθερή και πολύ σοβαρή αξιόπιστη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και των αρμόδιων αρχών και οργανισμών για αυτά τα προϊόντα παραχάραξης. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, παρόλο που ξέρουμε ότι είναι δύσκολα στην πράξη να πραγματοποιηθούν. Τώρα, όσον αφορά ένα σύστημα πιστοποίησης, ένα νέο ευρωπαϊκό σήμα πιστοποίησης, μέχρι τώρα δεν μπορούμε να πούμε ότι το ευρωπαϊκό σήμα μας ικανοποιεί. Βεβαίως δίνεται μια ένδειξη στον καταναλωτή Παρόλα αυτά, οι πληροφορίες που δίνονται από το Ευρωπαϊκό Σήμα δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε σήμερα εδώ. Εμείς προσπαθούμε να προστατεύσουμε περισσότερο τα ευρωπαϊκά πρότυπα, το Ευρωπαϊκό Σήμα. Βεβαίως υπάρχουν στις χώρες μέλη διαφορετικά συστήματα πτιστοποίησης. Από την άλλη μεριά υπάρχουν και οι παραποιήσεις ή ε, απομιμήσεις ε, ένα προϊόν πολύ χαμηλότερης ποιότητας το οποίο δεν πληρεί τα κριτήρια και τα πρότυπα ποιότητας, προστασίας και ασφάλειας μπορεί να έχει ένα σύστημα πιστοποίησης ή ένα σήμα το οποίο να είναι και αυτό απομίμηση. Παραδείγματος χάρη μια πετσέτα με το σήμα Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Καταλαβαίνετε ότι μια πετσέτα η οποία έχει το σήμα CE, Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ εμείς ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν θα έπρεπε να το έχει, αυτό ήδη είναι μια πράξη παραποίησης. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε τρόπους να μην υπάρχει καταχρηστική χρησιμοποίηση αυτού του σήματος και θα πρέπει να βρούμε τρόπους να αντιμετωπίσουμε αυτά τα φαινόμενα. Ένα σύστημα αποτελεσματικό στην ε, Αγγλία παραδείγματο χάρη και στις Ηνωμένε Πολιτείες υπάρχουν τέτοια συστήματα τα οποία όμως αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευρέως και εκτός των χωρών αυτών. Συζήτησα με πολλούς ε, για το θέμα αυτό και πιστεύω ότι το θέμα έχει οριμάσει και με πολύ μικρό κόστος και επιμένω σε αυτό μπορούμε να φτάσουμε σε ένα σύστημα αποτελεσματικό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι ίσως ε, μια προφορική ερώτηση ή έστω μια ακρόαση θα μπορούσε να μας βοηθήσει να εμβαθύνουμε στο θέμα αυτό. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι παρακολούθηση, έλεγχος της αγοράς. Και βεβαίως δεν έχω χρόνο αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μου, αλλά θέλω να σας πω ότι έχω οκτώ τροπολογίες οι οποίες θα διευρύνουν διάφορες πτυχές αυτής της ε, έκθεσης. Δεν μπορώ τώρα να σας τις παρουσιάσω όλες. Ελπίζω να μην ξέχασα κάτι σημαντικό σε αυτά που είπα. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Ρόιτοβα, λέει ο Πρόεδρος. Θέλω να υπενθυμίσω στα μέλη ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι την Παρασκευή 26 του μηνός το απόγευμα. Κοιτάξτε, θα σας δώσω το λόγο κύριε Ρέμπο, αλλά πρέπει να σας πω ότι δεν έχουμε πλέον χρόνο. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο. Αυτή η πολιτική η καινούργια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και τα όσα προετοιμάζονται τι μα συνέταξα. Ήταν κάπω βιαστικά, δεν διαθέτα και ούτε εγώ πολύ χρονικό διάστημα. Η Ήτρε αυτή η επιτροπή είχε αποφασίσει να εξετάσει αυτό το σχέδιο πολύ γρήγορα και θελήσαμε να γνωστοποιήσουμε και στην Επιτροπή την ε, άποψη του Κοινοβουλίου πριν ε, να δημοσιοποιήσει το πρόγραμμά της ε, καινοτομίας. Ε, κανονικά θα πρέπει να ολοκληρωθούν αυτά αυτή τη χρονιά, αλλά δεν ξέρω μήπως σημειωθούν και καθυστερήσεις. Σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής, βλέπουμε τις διάφορες πτυχές της καινοτομίας, των νέων στοιχείων, τις προκλήσεις και τα όσα παραμένουν για να πραγματοποιηθούν για την ανακοίνωση. Εδώ πρόκειται για μένα είδος εισαγωγή ε, στο όλο σχέδιο της Επιτροπής αργότερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Νομίζω ε, ότι προχωράει στον τομέα της καινοτομίας, αλλά παραμένουν άλλοι τα αρκετά προβλήματα. Κάτι που δεν είναι πια βέβαια βασικό πρόβλημα είναι εκείνο που έχει σχέση με τη γνώση. Από την άλλη μεριά θα πρέπει έγκαιρα ορισμένα πράγματα να εφαρμοστούν. Θα πρέπει η θεωρία να αποτελέσει στοιχείο πρακτικής εφαρμογής και να προωθήσουμε αυτά τα νέα προϊόντα. Έχουμε τις γνώσεις αλλά δεν γνωρίζουμε πώς περισσότερο κατάλληλα θα τις εφαρμόσουμε με την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ ανταγωνιζόμεθα και από πρακτικής πλευράς ε, το πρόβλημα το αντιμετωπίζουν οι εταιρείε, οι επιχειρήσεις και επίσης η διαχείριση της καινοτομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα ήθελα να τονίσω διάφορες πτυχές. Την ε, σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα πρέπει να προσέχουμε ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εργάζονται μέσα στις κατάλληλες συνθήκες για την όλη ανάπτυξη. Και δεν θα πρέπει να παρεμποδίζουμε την ανάπτυξη αυτή. Ε, διάφορες ρυθμίσεις ε, και ε, αυτές οι πιστοποίησεις ε, πάνω σε αυτά χρειάζεται επίσης να επαγρυπνούμε και το σύστημα της ε, άδεια καινοτομίας, ευρεσιτεχνίας είναι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό εδώ στην Ευρώπη αυτή την περίοδο, αυτή τη στιγμή. Και χρειάζεται, παραλαμβάνω, να επαγρυπνούμε πάνω σε αυτήν την τομέα και χρειάζεται να αλλάξουμε το όλο σύστημα. Χρειάζεται μια ευρωπαϊκή πιστοποίηση και συνόλφος εργάστηκε ιδιαίτερα πάνω σε αυτό αλλά χρειάζεται να πετύχουμε ακόμα αρκετά πράγματα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικές πτυχές επίσης για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί η συνθήκη της Λισαβόνας ε, μας ε, προσφέρει ορισμένες δυνατότητες και αρμοδιότητες και για τις πιστοποιήσεις αυτές ε, που αναφερόταν και στην όλη στην, στο όλο θέμα της συναπόφασης. Εδώ είναι πολύ σημαντικό να ε, μάθουμε πολλά και από τα όσα πετυχαίνουν οι Αμερικανοί στον τομέα αυτό. Χρειαζόμαστε περισσότερη ευκαμψία και ευληγησία σχετικά με την όλη διαχείριση της καινοτομίας στην Ευρώπη. Είναι ένα σύστημα που κοστίζει πάρα πολλά χρήματα. Χρειάζεται μια χρηματοδότηση και επίσης θα πρέπει να είναι κάπως πιο εύκαμπτη η όλη πρωτοβουλία αυτή στο σύνολό τη. Δεν μπορεί να περιμένουν ένα-δύο χρόνια οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να εφαρμοστούν αυτές οι καινοτομίες, δηλαδή από τη στιγμή που θα αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρηματοδοτήσει αυτές τις ενέργειες. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν διαθέτουν τόσα χρήματα και επίσης ε, στα πλαίσια της Επιτροπής η κατανομή αρμοδιοτήτων θα πρέπει να επανεξεταστεί γιατί ορισμένες πτυχές αυτής της πολιτικής ε, αντιμετωπίζονται από δύο διαφορετικά τμήματα. Χρειάζεται μια ομάδα περισσότερο ευλίγιστη και εύκαμπτη και ο κύριος Γκλίν ε, νομίζουμε ότι είναι πολύ καλή αυτή η ιδέα και ελπίζουμε και να εφαρμοστεί. Και χρειάζεται μια ευρύτερη έννοια της καινοτομίας. Δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για καινοτομία σε σχέση με την έρευνα. Χρειάζεται να μιλάμε και για την ζήτηση σε θέματα καινοτομίας που βασίζονται ακριβώς στις ανάγκες των πολιτών, στις ανάγκες της κοινωνίας μας. Από τη στιγμή που σημειώνεται μια ανάγκη. Εμείς μπορούμε ευκολότερα να προωθήσουμε ένα προϊόν που να περιέχει αυτά τα στοιχεία, τα καινοτόμα. Όσον αφορά τώρα τις τροπολογίες, διαθέτουμε δύο μέρες και για την κατάθεση των τροπολογιών αυτών, την υποβολή τους, γι' αυτό πρέπει να διηγήσουμε πολύ γρήγορα. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Κρόιτσμαν. Κυρία Ρούλε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, GT, μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση όσον αφορά την καινοτομία, όσον αφορά την απασχόληση, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Θα ήθελα όμως εδώ να πω ότι υπάρχουν ε, διαφορετικές ε, δομές που αφορούν το θέμα αυτό στην Επιτροπή και χρειάζεται καλύτερο συντονισμός. Όντως αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε στην Επιτροπή σε πολλά επίπεδα, διπλές ε, δομές. Όσον αφορά την καινοτομία, βεβαίω το θέμα αυτό έχει αρνητικέ συνέπειες. Βλέπουμε όμω ότι στη Γενική Διεύθυνση για την Εσωτερική Αγορά, όταν μιλάμε για καινοτομία παραδείγματο χάρη, βλέπουμε ότι η ιδέα της καινοτομίας είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι όμως κάτι που είναι συμπληρωματικό αν θέλετε. Δεν είναι η κεντρική ιδέα όπως θα έπρεπε να είναι. Αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση όσον αφορά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ σημαντικό να αποφύγουμε το γεγονός ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις υποφέρουν σήμερα. Οι μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες εποφελούνται από τις διαδικασίες αυτές οι οποίες είναι δύσκολες, βαριές και έχουν και ένα συγκεκριμένο κόστος. Το ίδιο ισχύει και για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας των λογισμικών, παραδείγματος χάνει. Οι μεγάλες επιχειρήσεις εποφελούνται, χρησιμοποιούν και οι μικρές υποφέρουν και δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σήμερα. Θα σε ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βάπολης πολύ σύντομα. Κύριε Πρόεδρε, ναι, πολύ σύντομα. Η κυρία Ρούλε είπε τα πιο σημαντικά σημεία τα οποία ήθελα και εγώ να θίξω. Η κυρία Ρούλε έχει εκφράσει κάποιες κριτικές που και εγώ ήθελα να εκφράσω εδώ. Αναρωτιέμαι λοιπόν, αυτός ο στόχος του 3% είναι κάτι που θα πρέπει να το διατηρήσουμε. Δηλαδή το 3% του επνοκρατών πρέπει να δίνεται στην έρευνα, στην καινοτομία. Μήπως πρέπει αυτό να φτάσει το 5% και εν πάση περιπτώσει να κάνουμε και μία αξιολόγηση του έχει γίνει μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ πολύ όμως και εγώ την εισηγήτρια. Thank you very uh, Ευχαριστούμε ε, κύριε Κρόιτσμαντ. Όσον αφορά τις... Ε, ε, παρατηρήσεις που έγιναν. Συμφωνώ και εγώ ε, με τα όσα είπαν οι προηγούμενοι. Αυτό το θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της βιώσιμης κατασκευής ε, μπορεί και αυτό μέσα από τις δημόσιες συμβάσεις να οδηγήσει σε καινοτόμα προϊόντα. Επίσης κάτι σημαντικό είναι η δημιουργία μιας κουλτούρας καινοτομίας. Φαίνεται ε, από την έκθεση ότι αναφέρεται και το θέμα νανοτεχνολογίας, βιοτεχνολογίας. Ας πούμε στην βιοτεχνολογία ο πρόεδρος Παρόζο έχει πει ότι πρόκειται για ένα θέμα που πρέπει να ρυθμίζεται εθνικά. Εγώ ήθελα να ρωτήσω ε, πώς μπορεί η Κομισιόν να συμβάλλει ώστε οι τεχνολογίες αυτές να έχουν μια ευκαιρία να μην είναι μόνο αυτοί που πιστεύουν στην καινοτομία που θα τις προωθούν, να θέλουμε μία κουλτούρα νέων τεχνολογιών. Γιατί χωρίς καινοτομία η Ευρώπη δεν θα έχει τη δυνατότητα να ε, εμπορεύεται τα προϊόντα της ε, στην παγκόσμια αγορά και η καινοτομία είναι η λέξη κλειδί για την ανταγωνιστικότητα της ε, ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Ευχαριστώ να σας θυμίσω ότι η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι Παρασκευή. ...26 το μεσημέρι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για τα σχόλια τους και όλα αυτά θα τα σωματώσω στην γνωμοδότησή μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τελειώνει το πρώτο κομμάτι της πρωινής συνεδρίασης και ε, παραχωρώ την έδρα.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 Πολύ καλά. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Να ευχαριστήσω στο σημείο αυτό όλα τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων που δέχτηκαν την πρόσκλησή μας αυτή και είναι μαζί μας για να συζητήσουμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα που είναι σημείο κλειδί για τα κράτη-μέλη και τις χώρες μας. Ε, έχει να κάνει με της, ε, με τα δικαιώματα των καταναλωτών θα δούμε τι σημαίνει αυτή η αντιπαράθεση, τι ακριβώς πιστεύουν, φρονούν τα κράτη-μέλη και τι γίνεται με τις προτάσεις των κρατών για να έχουν ένα πλήρη ρόλο και μια άποψη για όλα όσα έχουν να κάνουν με τα νομιμαδικαιώματα των καταναλωτών. Μετά από τη συνθήκη της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει περισσότερες αρμοδιότητες και δυνατότητα συναπόφασης με την Επιτροπή. Γι' αυτό αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το εργαλείο αυτό αντιπαραθέσεις να χρησιμοποιηθεί για να πετύχουμε νόμους χρήσιμους που να μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα στο εσωτερικό των κρατών μας σαν εισηγητής για τη σημαντική αυτή πτυχή, ο κύριος Βάμπ θα λάβει το λόγο και μετά θα λάβουν το λόγο οι ε, εθνικοί βουλευτές ε, και μετά έχουμε δύο ακριβώς που θα λάβουν το λόγο, δύο, ένας ευρωβουλευτής στη συνέχεια και μετά δύο βουλευτές από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Σας παρακαλώ αυτό το έντυπο συμπληρώστε το για να σας δοθεί και ο λόγος. Και έτσι λοιπόν θα ήθελα να σας πω τα δύο-τρία λεπτά να σεβαστείτε. Ε, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε διάλογο, να μπορέσουν να λάβουν το λόγο όσοι τον επιθυμούν και θα ήθελα να καλωσορίσω, να καλωσορίσω όλους, συγγνώμη και για την προφορά των ονομάτων τους, καλωσόρισαν, καλωσόρισε μάλλον ο κύριος Μπάτερλερ ή κάπως έτσι διστάζει η πρόεδρος, α, απόν θα έρθει σε λίγο. Το λόγο έχει ο κύριος Σβάμπ που θα μας γνωστοποιήσει διάφορες ιδέες του για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Ως εισηγητής ε, για τα δικαιώματα των καταναλωτών είναι μεγάλη μου χαρά ως εκπρόσωπος ε, ε, μαζί σας να συναλλαγώ σήμερα που είστε εδώ ως εκπρόσωποι των, των Εθνικών Κοινοβουλίων. Έχουμε σήμερα μια συγκεκριμένη πρόταση και σήμερα ε, συμφωνούμε στην Επιτροπή ότι δεν θέλουμε να ψηφίσουμε έτσι το κείμενο της Κομισιόν και θέλουμε, από όσα μας είπατε κι εσείς ε, με, τις τελευταίες σας ε, με την τελευταία συμβολή, να επηρεάσουμε αυτό το έγγραφο. Καταρχάς, να πω ότι η κατάσταση στην, στην Ευρωζώνη είναι κάτι που μας κάνει όλους να σπάμε το κεφάλι μας. Η διάδοση ε, ψευδών ε, δεδομένων να κάνει ακόμα πιο δύσκολη τη σημερινή κατάσταση. Για τις στατιστικές του 2008 ήμουν εισηγητής και θυμάμαι πολύ καλά ότι τότε οι κυβερνήσεις ζητούσαν να μην υπάρχει ε, τόσο αυστηρός έλεγχος από την Eurostat. Σήμερα βλέπουμε τις επιπτώσεις και θα ήταν καλύτερο εάν η έλεγχη ήδη τότε ήταν πιο ισχυρή από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ προσωπικά λοιπόν θεωρώ ότι σε κάποιες συζητήσεις στην Ευρώπη θα πρέπει να είμαστε πιο ειλικρινείς και πιο ρεαλιστές. Θα πρέπει να είναι δυνατή η Ευρώπη στα σωστά σημεία. Ειδικότερα όσον αφορά λοιπόν στην οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών, τους επόμενους μήνες θα έχουμε μία ανοιχτή συζήτηση και θα συζητήσουμε για τα πλεονεκτήματα, για τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και την εσωτερική αγορά γενικότερα με ανοιχτό τρόπο. Θέλουμε να βγάλουμε συμπεράσματα, όμως εξ αρχής πρέπει να έχουμε ε, καλή συζήτηση. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα ως εισηγητής να ε, διασφαλίσω ότι θα γίνουν αυτές οι συζητήσεις ε, με όλους τους ενδιαφερόμενους. Στις διαφουλεύσεις μας στην Επιτροπή τους τελευταίους μήνες συζητήσαμε κεφάλαιο προς κεφάλαιο και είδαμε ε, πώς ε, μπορούμε να ε, οριστικοποιήσουμε και κάποιες λεπτομέρειες πέρα από ομάδες κτλ. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι δεν θα γίνει μια πλήρης εναρμόνιση, αλλά ο στόχος αυτής της πλήρους εναρμόνισης πρέπει να προωθηθεί και να είναι ξεκάθαρη η στόχη. Στη σημερινή σας μας συναεδρίαση, με μία πρόταση για ένα έγγραφα εργασίας σας παρουσιάζω τα αποτελέσματα ε, αυτών των συζητήσεων για να μπορέσουμε να υιοθετήσουμε μαζί με σας αυτό το έγγραφο. Θεωρώ επίσης ε, ότι σήμερα η συζήτησή μας θα πρέπει να είναι το φαλτήριο. Σημαντική είναι η απλούστευση ε, του δικαίου των καταναλωτών, ε, ειδικότερα όσον αφορά το λιανικό εμπόριο ή ε, το εμπόριο εξ αποστάσεως. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλο και περισσότερο είναι σε απόσταση από τους ε, καταναλωτές τους. Έτσι, ε, παρόλο που υπάρχει αυτή η δυνατότητα, δεν είναι σωστό το εμποριο εξ αποστασεως οι μικρομεσαιες επιχειρησεις ολο και περισσοτερο ειναι σε αποσταση απο τους καταναλωτες τους ετσι παρολο που υπαρχει αυτη η δυνατοτητα δεν ειναι σωστο το πλαισιο και δεν εκμεταλλεύονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτές τις δυνατότητες και δαπανώνται πολλά ε, χρήματα για τις ε, συμβάσεις πώλησης. Αυτό είναι ένα φρένο στην ανάπτυξη και οδηγεί στη μη εκμετάλλευση του πολιτιστικού ε, και οικονομικού δυναμικού στην ΕΕ. Ευρώπη. Γι' αυτό είναι μεγάλη σημασία να έχουμε μια πλήρη εναρμόνιση για όλους τους καταναλωτές ε, σε επίπεδο αξιόπιστων ευρωπαϊκών στάνταρ. Πρέπει οι καταναλωτές να είναι σίγουροι ότι έχουν δικαίωμα επαναχώρησης, ε, ε, έχουν όλα τους τα δικαιώματα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι μπορούν να τα εφαρμόσουν. Επίσης, πρέπει να προσέξουμε ότι στο δίκαιο των καταναλωτών ε, θα πρέπει η προστασία των καταναλωτών σε ορισμένους τομείς ειδικότερα να έχει ε, υψηλό επίπεδο. Και γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε έξυπνες λύσεις για την εφαρμογή αυτής της πλήρους εναρμόνισης. Ε, στο πρώτο άρθρο της οδηγίας υπάρχουν, αναφέρεται η ανάγκη για βελτιώσεις σχετικά με τους ορισμούς. Κάποιοι ορισμοί δεν είναι ακριβείς και δεν δίνουν εγγύηση ότι χρησιμοποιούνται οι κατάλληλοι κανόνες για το κατάλληλο αντικείμενο. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να βαρύνονται με πολλές ε, υποχρεώσεις πληροφόρησης. Θα πρέπει όμως ταυτόχρονα να λαμβάνουν και τις απαραίτητες πληροφορίες οι καταναλωτές, να έχουν πληροφορίες για ποιότητα και όχι μόνο σε επίπεδο ποσότητας. Θεωρώ λοιπόν ότι ε, οι καταναλωτές θα μπορούν και μέσω ε, διαδικτυακών τόπων όπως το eBay να ε, συναλλάσσονται με ασφάλεια για τις ε, μικρομισές επιχειρήσεις για να μειωθούν οι νομικές ε, δαπάνες ε, θα πρέπει να υπάρχει ένα πρότυπο για το δικαίωμα υπαναχώρησης ώστε να υπάρχει ένας απλός τρόπος οι καταναλωτές να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και να έχουν ασφάλεια δικαίου. Για το κεφάλαιο 4 έχουν γίνει πολύ σοβαρές συζητήσεις και πολλοί βουλευτές ανέφεραν ότι ε, πολλά παραδοσιακά ε, δικαιώματα όπως το μπίσκασε και το Right to Reject θα πέσουν σε ε, δυνότερη θέση. Επίσης, ένα δεκαετές δικαίωμα διασφάλισης για τα προϊόντα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ε, άλλο ένα θέμα που ετέθη. Έτσι, η εναρμόνιση θεωρήθηκε ως η πιο έξυπνη λύση. Για να αποφύγουμε λοιπόν ε, τα προβλήματα, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι καταναλωτές είναι απλώς σε θέση να εφαρμόσουν τα δικαιώματά τους. Επίσης, μόνο μέσα στις ε, προθεσμίες θα μπορεί ένας καταναλωτής να χρησιμοποιήσει τα δικαιώματά του. Για το κεφάλαιο 5 να πω ότι ε, αναφέρθηκε ότι ε, μια μαύρη λύση, λίστα, συγγνώμη, η οποία θα πρέπει και αυτή να εναρμονιστεί. Είναι κάποιες ρήτρες που είναι ε, κοινός τόπος, για παράδειγμα, ε, η εναρμόνιση ε, των θεμάτων της ε, ευθύνης, εμπορικής ευθύνης. Αν αυτό μπορεί να γίνει βέβαια γενικά για τις ρήτρε, θα το εξετάσουμε. Θα πρέπει επίσης να διατηρηθεί ο δημοκρατικός έλεγχος έτσι ώστε ε, να ε, δούμε μέσα από τη διαδικασία της επιτροπολογίας τι θα γίνει με τις ε, περαιτέρω απαγορεύσεις. Θα πρέπει μετά το, τη Συνδίκη της Λισαβόνας η, η διαδικασία αυτή να αλλάξει. Αυτά θεωρώ λοιπόν ότι είναι η βάση για τη σημερινή μας συζήτηση. Η Επιτροπή μας θέλει να δουλέψει για βελτίωση ε, της εργασίας σε αυτόν τον τομέα, ειδικότερα για ένα κοινό πλώσιο, πλαίσιο εργασίας. Και θα πρέπει να, έχουμε υπόψη μας και το κοινοτικό και εκτιμένο. Θεωρώ ότι θα βελτιωθεί το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα γίνουμε πιο ισχυρές επιχειρήσεις. Θα έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης. Ελπίζω ότι η κρίση θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί για να αυξηθεί και η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην αγορά. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Πολύ καλά. Τον κύριο Σουφάλμπε θα θέλαμε να τον ευχαριστήσουμε για την εισήγησή του αυτή και οι βουλευτές από τα Εθνικά Κοινοβούλια έχουν το λόγο. Επιθυμούμε να ακούσουμε τις απόψεις, τις απόψεις τους. Καραμανλή. Όχι, συγγνώμη, συγγνώμη, ναι. Από το Γαλλικό Κοινοβούλιο και με βιντεοδιάσκεψη όπως είχε προσδευθεί. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, με ιδιαίτερη προσοχή άκουσα την παρέμβαση του κύριου Σφάλμπ και ασχολούμεθα με την οδηγία αυτή εδώ και κάπως χρονικό διάστημα. Όλοι μας εθνικοί βουλευτές και ευρωβουλευτές συμφωνούμε και συμμεριζόμαστε τις ίδιες ανησυχίες πέρα από τις πολιτικές μας ε, πεπιθήσεις. Ε, είμαστε εκλεγμένοι από το λαό και είμαστε και πεπισμένοι ότι θα πρέπει να μεταβληθεί το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2008 και αυτό απαιτείται ακόμη περισσότερο με την οικονομική κρίση και περισσότερες ανησυχίες εκφράζονται από τους πολίτες μας τώρα. Χρειάζεται υψηλή προστασία του καταναλωτού όπως ε, λέει και η συνθήκη της Αβώνας. Δεν είναι μόνο νομικό αλλά κοινωνικό και οικονομικό σαν επιταγή και ακριβώς και μέσω της Αθαγένειας και με το κοινό μας κοινωνικό πρότυπο και νομίζω ότι πρόκειται και για κάτι προστατευτικό για εκείνους που αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα. Ε, τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει και μια δυσπιστία απέναντι στις τράπεζες και πρέπει να αποφεύγουμε οτιδήποτε μπορεί να αποσταθεροποιήσει τον καταναλωτή και την πιστοσύνη του. Και ακριβώς ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το Γαλλικό Κοινοβούλιο, αφιέρωσε τρεις συναντήσεις ε, στην οδηγία με βιοδιάσκεψη 22 Ιανίου που μας πέρασε. Πρώτη φορά έγινε αυτό μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι λέμε ότι με τον τρόπο αυτό θα πρέπει να συνεχίσουμε τις ανταλλαγές απόψεων με, ανάμεσα στα Εθνικά Κοινοβούλια και είχαμε πρώτα απ' όλα ομόφωνα τη, ε, Νοέμβριο που μας πέρασε ότι όλα αυτά θα πρέπει να συμπληρωθούν και παρακολουθούμε την εξέλιξη του θέματος τους τέσσερις προσανατολισμούς και γενικές κατευθύνσεις προτάθηκα να υπενθυμίσω όχι οπισθοδρόμηση όσον αφορά την προστασία του καλωτού ένα κείμενο που να αφορά τα κύρια σημεία και για την επικουρικότητα και με τις αρμόδιότητες πάντα των κρατών μελών έχουν και επίσης μια στόχευση για τις ρυθμίσεις εκείνες που απαιτείται μόνο. Επίσης, πεδίο εφαρμογή και απέναντι στο ευρωπαϊκό δίκαιο και στο εθνικό δίκαιο, το θα πρέπει να, πρέπει να παραμείνει σε ισχύ, το αστικό δίκαιο κυρίω και να επενθυμίσουμε ότι είχαμε ένα πρώτο ε, κείμενο αυτού του προσεχούς κοινού και με τη δυνατότητα με περαιτέρω προστασίας και σε άλλες κατηγορίες επαγγελματικές, άλλους κλάδους και γενική ενημέρωση για το τι διακυβεύεται εκεί στην εσωτερική αγορά κλπ. Και, και τις συναλλαγές και τις συμφωνίες ε, και να ισχύουν όλα αυτά πέρα από εκεί που αφορά η αγορά και επίσης εγγύηση μια κάποια ευκαμψία και ευληγησία για την ε, επιλογή και ειδικού μηχανισμούς που ισχύουν σε ορισμένα κράτη όπως επανσχάριστα ε, κρυφά ελαττώματα των διαφόρων προϊόντων. Όλα αυτά, σε αυτά, εξετάσαμε και τη διάρκεια των συνομιλίων μας. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρεύουσα. Θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω και δύο μέλη του Νορβηγικού Κοινοβουλίου, Σίμενσεν και Άνσεν. Βρίσκονται ανάμεσά μας και παρακολουθούν τη συζήτησή μας από το Νορβηγικό λοιπόν Κοινοβούλιο. Για το θέμα αυτό και πάλι, ο γερουσιαστής Κάζολη από, το, από την γερουσία την Ιταλική. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ. Θέλω να σε ευαισθητοποιήσω για ορισμένε ειδικέ πτυχέ τη οδηγία αυτή για την προστασία του καταναλωτού. Αυτό που φαίνεται στα πλαίσια των εργασιών του Συμβουλίου για την επέκταση σε 10 χρόνια της νόμιμης εγγύησης των που προσφέρεται από τους πολίτες και απαιτείται ακριβώς εξειδίκευση αυτών των κατηγοριών τι αφορά και με μια επέκταση της εγγύησης και αυτό είναι ισόφελος του καταναλωτού και στο μέλλον και θα πρέπει ίσως να είναι όμως και ένα διαβατήριο για τα διάφορα προϊόντα και τι γίνεται αν το πάνε μέχρι 9,5 χρόνια μόνο και τι γίνεται ανάμεσα σε καταναλωτή και πολιτή πέρα από τα δύο χρόνια χωρίς να συμμετέχει ο ίδιος ο παραγωγός. Ε, για τα προϊόντα αυτά χρειάζεται να συμφωνήσουμε όλοι ότι η βιομηχανία θα πρέπει να καταβάλει προσπάθεια για να βελτιώσει τις υπηρεσίες της ε, στον καταναλωτή και δεν θα έπρεπε να υποχρώνουμε τις εταιρείε να καλύπτουν τα προϊόντα για 5-10 χρόνια. Ε, χρειάζεται να δούμε ακριβώ τα πρέπει να κάνουμε και ο καταναλωτή θα μπορούσε να διαλέξει αν το επιθυμεί αυτό ή όχι. Και σύμφωνα και με την προσφορά υπηρεσιών ε, για ένα σέρβις, ε, για περισσότερη μακρύτερη ζωή στον, ε, στα προϊόντα όπως ακριβώς γίνεται και με τα αυτοκίνητα πέρα από το κοινό όνομα εγγύηση, θα πρέπει να γίνεται μια εξήγηση αυτών που εμπεριέχει για τη διάρκεια του προϊόντος και έτσι ο καταναλωτής να έχει την καλύτερη δυνατή προστασία. Τελευταίο σημείο που έχει να κάνει για το τρίτο εδάφιο της κειμένου οδηγίας ε, και για τις πληροφορίες για τους καταναλωτές και η επιστροφή για τα συμβόλαια που κλείνονται από απόσταση και τις υποχρεώσεις των διαφόρων εάν εφαρμοστούν όλα αυτά για τη μεταφορά ας πούμε την ε, στερομική θα πρέπει να ισχύσει πάντα και το δικαίωμα άρνησης, ακύρωσης, κάτι που δεν θα πρέπει να θίξει τους καταναλωτές. Οι διάφορες ε, εταιρείε ε, μεταφορών ε, θα είχαν όμως μεγάλες ζημιές και ουσιαστικά θα είχαν λιγότερο θετικές προσφόρες προς τους καταναλωτές μέσω υψηλότερης τιμής εισιτηρίου. Ευχαριστούμε τον Γερουσιαστή, λέει η και τώρα Γκέπαρντα σκιώδης συσυγήτρια για την οδηγία αυτή. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν σας ευχαριστώ για αυτή τη συνάντηση. Είναι εξαιρετικά σημαντικό όχι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και οι συνάδελφοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια να μπορούν ε, καθώς και τα μέλη των διαφόρων ε, γερουσιών, ε, βουλών, αλλά και από το γερμανικό Bundesrat, να μπορέσουν να συμμετάσχουν σε αυτή τη συζήτηση. Η προστασία των ε, καταναλωτών δεν είναι απλώς μια υπηρεσία που προσφέρουμε. Προσφέρουμε δικαιώματα και προσφέρουμε και μια ασφάλεια στους Ευρωπαίους πολίτες. Και αυτό είναι και το νόημα αυτής της προσπάθειας. Γι' αυτό ακριβώς και θέλουμε να διατηρήσουμε αυτή την αρμοδιότητα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σκοπός μας δεν είναι να δημιουργήσουμε μια μεγάλη εσωτερική αγορά χωρίς να προσφέρουμε απολύτως καμία προστασία στους Ευρωπαίους καταναλωτές. Ακούστηκε καταρχήν η ιδέα ότι η πλήρης εναρμόνιση δεν είναι η σωστή κατεύθυνση την οποία θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Υπάρχει η ιδέα της ελάχιστης ε, εναρμόνισης όσον αφορά την ε, προστασία των καταναλωτών και το θέμα που μας απασχολεί μας εδώ είναι να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε με ορισμούς, παραδείγματος χάρη, όσον αφορά την ε, επιστροφή, της αποζημιώσεις. Υπάρχουν τομείς με πάρα πολλές δυσκολίες γιατί η προστασία του καταναλωτή όταν παραδείγματο χάρη μιλάμε για ελάχιστη εναρμόνιση αντιμετωπίζουμε σήμερα προβλήματα διαφορετικής ερμηνείας, διαφορετικών ορισμών από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Να μην ξεχνάμε λοιπόν ότι ξεκινάμε από διαφορετικές ε, ε, καταστάσεις από διαφορετικά σημεία κίνηση στο κάθε κρατος μέλος και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το σεβαστούμε. Τώρα, οι οργανώσεις των καταναλωτών παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στα κράτη-μέλη με διαφορετικό επίπεδο συμμετοχής στις κοινωνίες των κρατών μελών και με διαφορετική παράδοση και ιστορικό ρόλο. Όταν όμως σήμερα βλέπουμε ότι υπάρχουν νέες προτάσεις, νέες ιδέες, νέες λύσεις, αυτές θα πρέπει να διαδίδονται στην Ευρώπη. Και εδώ βλέπουμε ότι το ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ακόμα ένα επίπεδο που δεν λειτουργεί ικανοποιητικά. Είναι αργό, οι νέες ιδέες δεν προχωρούν, γι' αυτό και θα ήθελα εδώ να ζητήσω από τις οργανώσεις των καταναλωτών, από τους αρμόδιους οργανισμού σε εθνικό επίπεδο να αναλάβουν αυτόν τον ρόλο. Η πλήρης εναρμόνιση δεν πρέπει να γίνει πραγματικότητα. Θέλουμε μια υπεύθυνη εναρμόνιση στους τομείς αυτούς όπου αυτό θα προσθέσει κάτι το θετικό. Τρίτο σημείο που θα ήθελα να υπογραμμίσω. Η πλήρης εναρμόνιση η οποία είναι αντίθετη αν θέλετε με μια στοχευμένη και συγκεκριμένη εναρμόνιση, είναι κάτι που το αντιμετωπίσαμε επίσης και με την οδηγία για την καταναλωτική πίστη. Εκεί είδαμε ακριβώς τα προβλήματα αυτής της ιδέας της πλήρους εναρμόνισης. Στο τέλος βλέπουμε ότι το περιβάλλον που δημιουργείται από μια τέτοια προσπάθεια πλήρους εναρμόνισης είναι ένα περιβάλλον με πολλά κενά, ανομοιογενές, χωρίς ευελιξία. Ακριβώς αυτό θέλω να πω σήμερα εδώ. Πρέπει να είμαστε βεβαίως προσεκτικοί, να προχωρήσουμε σταδιακά, άρθρο προς άρθρο. Κύριε Σφάμπ, αναφέρατε πολλά ε, παραδείγματα. Παραδείγματο χάρη, οι εγγύσει, οι αποζημιώσει, το δικαίωμα επιστροφής, υποχώρηση, όλα αυτά βεβαίω θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε λαμβάνοντας υπόψη μας ποιο είναι το πιο υψηλό επίπεδο προστασίας στην κάθε χώρα. Αυτό θα ήταν το ιδανικό αν θέλετε. Αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και πρέπει να επαναλάβουμε τη βασική ιδέα που διδαχτήκαμε από τη μέχρι τώρα εμπειρία μας, η ελάχιστη εναρμόνιση, η εναρμόνιση η στοχευμένη. Αυτός είναι ο σωστός δρόμος, η σωστή κατεύθυνση, έτσι ώστε οι καταναλωτές να αποκτήσουν περισσότερη εμπιστοσύνη στην κοινωτική πολιτική. Ευχαριστούμε την κυρία Γκέπαρν. Παρακαλώ, σεβαστείτε το χρόνο ομιλίας. Έχουμε πάρα πολλούς που επιθυμούν να λάβουν το λόγο και γι' αυτό δύο-τρία λεπτά ο καθένας σας. Παρακαλώ στους εθνικούς βουλευτές. Γκόμπερ από το Γαλλικό Κοινοβούλιο. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Μετά από όσα είπε η κυρία Καραμαλή που είναι εισηγήτρια στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο Γαλλικό Κοινοβούλιο να προσθέσω μερικά πράγματα και να κερδίσω και κάποιο χρόνο. Όσον αφορά την αρχή, δύο προσεγγίσει ε, για την κατανάλωση, για εσωτερική αγορά και προστασία των καταναλωτών δεν είναι αντιφατικά αυτά τα δύο, είναι συμπληρωματικά. Και θα θέλουμε μια καλύτερη ισορροπία και επίση, το μελλοντικό κείμενο δεν θα πρέπει να είναι μια πιστοδρόμηση αφορά την προστασία του καταναλωτή. Αυτό να μην υπάρχει έτσι ε, αφαίρεση στοιχείων μα ισχύουν τώρα που είναι ελάχιστη εφαρμογή απέναντι στα εθνικά δικαία και η πλήρη εναρμόνιση όπω η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προβλέπει ε, σημαίνει ιδιαίτερα απειλή κυρίω για τον καταναλωτή. Γι' αυτό να είμαστε προσεκτικοί και ο ίδιος ο καταναλωτής θα πρέπει να δει ακριβώς αν είναι μια ψευδρόμηση μια πρόοδος και όλοι μας το έχουμε δει και σε περιπτώσεις αντιπαράθεσης όταν δεν έχουμε απαραίτητα στοιχεία και να ξέρουμε πότε μπορούμε να οπισθοχωρήσουμε και όχι μόνο πότε μπορούμε να προχωρήσουμε. Εδώ δεν θα πρέπει να απαγορεύουμε στα κράτη-μέλη να παρεμβαίνουν να χρειάζεται όταν υπάρχει μια ειδική δυσκολία και καταρχή είναι ακριβώς ε, η εθνική πλευρά που θα πρέπει να φασίσει πάνω σε αυτά και ορισμένα πράγματα που δεν αντιμετωπίζει ποτέ τη οδηγία, αλλά θα ήταν καλό να έχουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων ε, ε, τα ψηφιακά προϊόντα και από τη στιγμή που δεν είναι σύμφωνα με τις ρυθμίσεις ε, και εάν ε, το μηχάνημα που τα διαβάζει δεν είναι το κατάλληλο και θα πρέπει, θα πρέπει να δούμε το δικαίωμα ακριβώ συμβολέου και το 28-8 δικαίωμα ακριβώ που να είναι συμπληρωματικό από εθνικής πλευράς και οι ομαδικές επίσης ενέργειες σε περίπτωση προβλήματος. Ευχαριστώ. Πολύ καλά, σας ευχαριστώ και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Ντέμεκ από, Αυστρία, από την Αυστριακή Γερουσία. Καλημέρα σας. Η άποψη της Αυστρίας, καταρχήν ε, και εδώ θα συμφωνήσω με τους προηγούμενους ομιλητές, είμαστε κατά της πλήρους εναρμόνισης. Θεωρούμε πραγματικά ότι αυτό θα ήταν ένα βήμα προς τα πίσω. Κοιτώντας το τι συμβαίνει στις ε, άλλες χώρες, θεωρούμε ότι στη χώρα μας έχουμε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή. Αυτό όμως που είναι ενδιαφέρον όταν μιλάμε για προστασία του καταναλωτή είναι ενδιαφέρον στις περιπτώσεις διαφορών, διαμάχης μεταξύ του καταναλωτή και του κόσμου των επιχειρήσεων. Μας ενδιαφέρει λοιπόν πραγματικά να διατηρήσουμε το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας στα διάφορα κράτη-μέλη και ως προς το περιεχόμενο αυτής της οδηγίας βεβαίως και θα πρέπει να υπάρξει ένα νομικό πλαίσιο υπάρχουν σημεία λοιπόν τα οποία θεωρούμε ενδιαφέροντα όσον αφορά παραδείγματο χάνει τις διάφορες διατάξεις για τη δυνατότητα αλλαγής γνώμης, οπισθοχώρησης, επιστροφής, της προθεσμίας, Επίσης, όσον αφορά τις διατάξεις για το συμβατικό δίκαιο, πιστεύω ότι εδώ πρέπει να παραμείνει ένα περιθώριο ελιγμού. Στη Γερμανία και στην Αυστρία, παραδείγματο χάρη, δεν μπορούμε να δεχτούμε 100% το αγγλοσαξονικό πνεύμα όσον αφορά τις, το συμβατικό δίκαιο. Και θεωρώ ότι, εν πάση περιπτώσει, το γενικό πνεύμα αυτής της προσπάθεια θα πρέπει να είναι όχι πλήρης αναρμόνιση και ύψιστη προστασία ανάλογα με την παράδοση της κάθε χώρα. Ευχαριστούμε τον γερουσιαστή Κρότμαν τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι από ό,τι άκουσα από όλου όσου πήραν το λόγο ότι δεν έχει νόημα εδώ η πλήρης αναρμόνιση σε κανένα τομέα καθότι όπως είπε και ο εισηγητής υπάρχουν διαφορετικές παραδόσεις και νοοτροπίες. Τελείως διαφορετικά αντιμετωπίζουν οι περιοχές, ε, τα γερμανικά κρατήδια, η Γερμανική Ομοσπονδία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν μέσα στη Γερμανία έχουμε τέτοιου είδους διαφορετικές προσεγγίσεις, τι θα γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μου αρέσει πολύ η έννοια της στοχευμένης εναρμόνισης, όπως είπε η κυρία Γκέπχαρτ. Ο ορισμός βεβαίως της εναρμόνισης, εκεί που αυτό είναι κάτι που προσθέτει, που βελτιώνει την κατάσταση. Είναι όπως η αρχή της επικουρικότητας. Θα κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό που κάνουμε καλύτερα από το τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό. Στην Ευρώπη όμως θα πρέπει να έχουμε ένα επίπεδο, ένα ελάχιστο επίπεδο και από εκεί και πέρα, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές παραδόσεις και θα πρέπει βεβαίως το ευρωπαϊκό επίπεδο να είναι γνωστό, να είναι γνωστό σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το αυστριακό παράδειγμα ήταν πολύ σωστό. Εκεί λοιπόν που μπορούμε να προχωρήσουμε στην εναρμόνιση, ναι. Ε, εκεί όμως που υπάρχει πολύ ψηλή προστασία, παραδείγματος χάνει σε ένα ε, συγκεκριμένο κράτος, αυτό θα πρέπει να το αφήσουμε. Κύριε Σφάμπ, έχετε δίκιο όταν λέτε ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε γενικές έννοιες, αρχές ευρωπαϊκές. Και αυτό βεβαίως σε τομείς που εξορισμού ξεπερνούν τα σύνορα και τα όρια, όπως παραδείγματος χάρη τα ηλεκτρονικά προϊόντα. Εκεί καταλαβαίνετε ότι σήμερα υπάρχει κενό. Υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν ε, και θα είναι σημαντική η συνεισφορά μας αν καταφέρουμε στον τομέα του διαδικτύου παραδείγματο χάρη να επιβάλλουμε ένα τέτοιο επίπεδο προστασίας Κάτι το οποίο είναι πολύ πιο δύσκολο από ότι στα υλικά προϊόντα, στι ηλεκτρικέ συσκευέ παραδείγματο χάρη, που είναι πιο εύκολο να επιβάλλουμε υψηλό επίπεδο προστασία. Ευχαριστούμε. Τακ, Γερμανό Υπουργό. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, και εγώ αναφέρω κάποιες θέσεις ως Πρόεδρος ε, της ε, Γερμανικής ε, Διάσκεψης Υπουργών για την Προστασία των ε, καταναλωτών. Θα σας δώσω την θέση του Bundesrat. Συμφωνώ ε, και με τα όσα είπε η κυρία Γκέρπραρτ. Το Bundesrat, ε, η Υπουργός Προστασίας των Καταναλωτών, έχουμε ως τώρα συμφωνήσει σε σχέση με την γνωμοδότηση που θα δώσουμε για αυτήν την οδηγία. Να υπογραμμίσω ότι μία πλήρης εναρμόνιση ε, σε τεχνικές λεπτομέρειες, για παράδειγμα, όσον αφορά στις ε, προθεσμίες, ε, θα ήταν λογική, αλλά όχι σε όλο το δίκαιο των καταναλωτών. Αυτό ήδη έχει υποθεί. Για μια τέτοια εναρμόνιση έχουμε ε, δεν έχουμε επαρκή βάση νομική και αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε. Υπάρχουν κρίσιμα σημεία, προτάσεις ε, για μια πολιτική καλύτερης ε, νομικής βάσης. Επίσης, όσον αφορά τα διάφορα κράτη-μελή και το επίπεδο το οποίο έχουν μέχρι τώρα, η κατάργηση αυτών των διαφορών θεωρούμε ότι θα ήταν εσφαλμένη. Όσον αφορά το ελάχιστο επίπεδο, Θεωρούμε βεβαίως ότι η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην νομοθεσία που έχει σαν σκοπό την προστασία των καταναλωτών είναι κάτι που σε αυτό θα πρέπει να ενδυναμωθεί και αυτό με πολύ συγκεκριμένα μέτρα καθώς και με την εξάλληψη των προβλημάτων που συνεχίζουν να υπάρχουν. Είναι επίσης πολύ σημαντικό και αυτό το έχουμε αναλάβει και επεξεργαστεί στην Γερμανία να αντιμετωπίσουμε τομείς ε, όπως αυτό της ε, ε, παράνομης διαφήμισης μέσω της, των τηλεπικοινωνιών και μέσω του διαδικτύου. Η απάντηση που μονίμως δίνουμε όταν προκύπτουν τέτοια προβλήματα είναι περιμένετε. Το ευρωπαϊκό επίπεδο είναι αρμόδιο. Την ίδια ώρα όμως βλέπουμε ότι τέτοιες καταχρηστικές πρακτικές καθώς και απάτες συνεχίζουν να λαμβάνουν χώρα και αυτό που τελειώνοντας θα ήθελα να πω είναι ότι πραγματικά στις νέες ρυθμίσεις που προσπαθούμε να επιβάλλουμε στην εσωτερική αγορά η προστασία του καταναλωτή θα πρέπει να είναι πολύ συγκεντρημένη να αποφευθούν και εργοστοκοπικές δραστηριότητες και να είμαστε διατεθειμένοι να αναλάβουμε αυτέ τι πρωτοβουλίε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προστασία του καταναλωτή. Σας ευχαριστώ πολύ γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μέχρι τώρα. Σα ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχει ο σκιώδη βασιλιστή του Ρούνεν, αν προφέρω καλά το όνομα, με συγχωρείτε λέει η πρόεδρο. Η κυρία. Ναι, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ είμαι εξ ονόματος, ακριβώς είμαι με τη διότητα μου σαν σκιώδης εισηγήτρια και είμαι υπέρ αυτής της εξέλιξης της οδηγίας με περισσότερη εμπιστοσύνη έτσι στην εσωτερική αγορά. Πρόκειται για μια βελτίωση της νομοθεσίας, δεν έχουμε καμία αντίρρηση πάνω σε όλα αυτά. Αλλά ανησυχούμε για κάτι ανησυχούμε για την πρόταση της Επιτροπής. Κριτική να ασκήσουμε σε δύο σημεία. Πρώτα απ' όλα, μια τυφλή, ας το πούμε έτσι, εναρμόνιση με νομικές συνέπειες και με πολλές αβεβαιότητες για τον καταναλωτή και μάλιστα σε κάθε γωνιά της Ευρώπης. Δεύτερο σημείο που θέλουμε να ασκήσουμε κριτική. Δεν βλέπουμε το τι δυνατότητες μπορούμε να εκμεταλλευτούμε. Θέλουμε μία... Βλέπουμε τι γίνεται ακριβώς ε, μια επικεντρωμένη εναρμόνιση εκεί που έχει νόημα αυτό και θέλουμε μια κάποια σαφήνεια νομική. Κάτι που μπορεί να γίνει, αν δούμε κατάλληλα το επίπεδο εναρμόνισης, είναι υπάρξει και μια εγγύηση για το μέλλον με περισσότερες ε, ε, ανάγκες και δυνατότητες για το μέλλον είναι όμως μια σημαντική θετική εξέλιξη. Νομίζω ότι έτσι μπορούμε να πετύχουμε κάτι τέτοιο ιδιαίτερα θετικό. Ευχαριστώ, λέει και η Πρόεδρος. Ε, δεν έχω στον καταλογό μου κανένα άλλο μιλητή από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Άρα λοιπόν οι Ευρωβουλευτές θα μπορούσαν να λάβουν το λόγο τώρα. Κάποιο άλλος να ρωτήσει για τελευταία φορά από Εθνικό Κοινοβούλιο. Όχι, κανείς. Ροϊτόα. Πασαρέλα, Ευχαριστώ πολύ. Να πω ότι έγινε τεράστια πρόοδος και να ευχαριστήσω τον συνάδελφο τον κύριο Σφάπο που μπόρεσε να ταυτοποιήσει τα προβλήματα που πρέπει να επιληθούν. Είναι πολύ σημαντικό να μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα και να υπάρχει ένα όραμα σχετικά με το πού θέλουμε να πάμε ε, αφού εγκρίνουμε αυτή την ε, οδηγία. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε ανταλλαγή απόψε με τα εθνικά κοινοβούλια. Αυτό το εγχείρημα είναι μακροπρόθεσμο και θα πρέπει να διαχωριστεί σε δύο φάσεις. Πρώτον, να ορίσουμε όρους, τους ορισμούς ε, που θα μας βοηθήσουν και εφόσον γίνει αυτό θα πρέπει να εναρμονίσουμε τα στάνταρτ. είναι σόφρον να κατανοούν και οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις τα minimum standard και αν είναι δυνατόν μετά να προχωρήσουμε και να αυξήσουμε αυτά τα πρότυπα. Γιατί σε πολλά ε, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτά είναι σε ψηλότερο επίπεδο από ό,τι σε άλλα. Εκεί που είναι σε ψηλότερο επίπεδο, στη δεύτερη φάση θα μπορέσουμε να συγχωνεύσουμε με υφιστάμενα στάνταρτ. Και αυτό είναι σημαντικό και για τις επιχειρήσεις και για τους καταναλωτές. Είναι σημαντικό να έχουν πληροφόρηση. Αυτή τη στιγμή όμως πρέπει καταρχάς να βρούμε τις διαφορές μεταξύ των στάνταρ που υπάρχουν στα διάφορα κράτη-μέλη. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν κάποιες, κάποια πρότυπα για τις εγγύησεις. Εμείς μπορούμε να τα εφαρμόσουμε ή θα ήταν μεγάλο το κόστος. θα ήταν καλό για τους καταναλωτές σε άλλα κράτη-μέλη. Αυτές οι διαφορές λοιπόν πρέπει να ε, ταυτοποιηθούν. Να πω τώρα στους εκπροσώπους από τη Γερμανία. Έχουμε τον κύριο Σφάπες και τις ηγητές και ανθρώπους από τον Bundestag της Γερμανίας. Η Γερμανία συνορεύει με πολλές χώρες αλλά τα στάνταρτ στην Γερμανία είναι συγκρίσιμα με αυτά που υπάρχουν στις ε, περιβάλλουσες χώρες, στις γειτονικές χώρες, Πολωνία, Γαλλία κτλ. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δικών σας προτύπων και των προτύπων που εφαρμόζουν οι γειτονικές χώρες. Μπορούμε και εμείς να έχουμε πληροφορίες σχετικά με αυτό μέσα από κάποιο website, κάποιο επίσημο σύνδεσμο, από κάποιο συνδέσμο προστασία των καταναλωτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μπορούν οι καταναλωτές από τις γειτονικές χώρες αν η προστασία στη Γερμανία είναι υψηλότερη ή πρέπει να, ε, έχουν, να βασίζονται στην προστασία που έχουν στην πατρίδα τους. Με συγχωρείτε, καθυστέρησα περιμένοντας ε, τις τελευταίες φράσεις της Γερμανίας. Η κυρία Ράφτη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Σουάπ για την εργασία που κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό με πάρα πολύ επιμέλεια. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμη η συζήτηση με τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Και αυτό όχι μόνο για να πάρουμε ιδέες, αλλά και για ένα πραγματικό δεδομένο που υπάρχει. Το πραγματικό δεδομένο είναι ότι ξεκινάμε από διαφορετικές εθνικές αφετηρίες έχω στο μυαλό μου την Ελλάδα από την οποία προέρχομαι, στην οποία θα έλεγα ότι έχουμε υψηλότερα δικαιώματα σε στους καταναλωτές σε σχέση με τα προτινόμενα από την οδηγία. Έτσι λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι όταν μιλάω έχω στο μυαλό μου το πώς μπορούν οι καταναλωτές να ωφεληθούν περισσότερο, κάτι που νομίζω ότι είναι στο μυαλό όλων. Άρα εκ των πραγμάτων αισθάνομαι ότι η πλήρης εναρμόνιση που δεν μας πηγαίνει στο υψηλότερο σημείο αλλά στο χαμηλότερο δεν είναι προς όφελος των καταναλωτών. Ε, θα θυμίσω εδώ ότι έχει ασχοληθεί και η Ελληνική Βουλή με το θέμα αυτό και έχει καταλήξει σε κάποια κοινά συμπεράσματα. Σε συμπεράσματα που λένε ε, ότι ουσιαστικά ε, θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει τον όρο ότι παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας μέσα από το σκεπτικό για μια πλήρη εναρμόνιση. Ε, απ' την άλλη πλευρά ε, θα έλεγα ότι έχοντας πάντοτε στο μυαλό μας τα συμφέροντα των καταναλωτών είναι πάρα πολύ εύστοχες οι παρατηρήσεις και οι ορισμοί που χρησιμοποίησε η κυρία Γκέπχαρτ κάθε ένας από αυτούς τους χαρακτηρισμούς έχει πίσω του ένα τεράστιο περιεχόμενο. Η υπεύθυνη εναρμόνιση. Η λέξη υπεύθυνη δεν είναι μόνο ένας επιθετικός προσδιορισμός που μπορεί να ακούγεται ευχάριστα και να προσφέρει ισορροπία στην κουβέντα. Είναι ένας χαρακτηρισμός που έχει να κάνει με την ευθύνη η ευθύνη πηγαίνει στο κράτος μέλος ή πηγαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήπως πηγαίνει και στις δύο πλευρές. Και αν πηγαίνει και στις δύο πλευρές όπως έτσι πρέπει να είναι, τι ποσοστό πρέπει να αναλογεί στην καθεμία. Είπε κάτι άλλο η Εύελιν Γκέπχαρτ. Στοχευμένη εναρμόνιση. Και εδώ η λέξη στοχευμένη έχει τεράστιο περιεχόμενο. Έρχεται στο μυαλό μου το διαδίκτυο. Είναι ένας στόχος πάρα πολύ συγκεκριμένος και ένας στόχος που θα τον βρίσκουμε συνεχώς στο μέλλον. Νομίζω ότι θα ίσως, ίσως να σκεφτούμε κάποια ξεχωριστά, κάποιες ξεχωριστές ρήτρες σε σχέση με τα δικαιώματα των καταναλωτών μέσα στο διαδίκτυο. Ε, υπάρχουν όπως αντιλαμβάνεστε και σκέπτομαι ότι έχει στο μυαλό το καθένας πάρα πολύ ξεχωριστοί τέτοιου είδους στόχοι που πρέπει να τους λάβουμε υπόψη. Ε, καταλήγοντας, για να σεβαστώ και το τρίλεπτο, ε, θα έλεγα ότι ο στόχος είναι η χρυσή ισορροπία. Ε, ξέρω ότι όσο εύκολο ακούγεται, τόσο δύσκολο είναι να επιτευχθεί. Αλλά έχω εμπιστοσύνη και στην Επιτροπή, έχω εμπιστοσύνη στο Κοινοβούλιο και έχω εμπιστοσύνη και στον κύριο Σουάμπ που κάνει τόσο διεξοδική εργασία. Ε, εκφράζοντας αυτή μου την εμπιστοσύνη, θέλω να πιστέψω ότι παράλληλα τον δεσμεύω για να κάνει το καλύτερο δυνατό στο πλαίσιο που εργαζόμαστε πάντα για τους καταναλωτές. Σας ευχαριστώ. Θα θέλαμε να σε ευχαριστήσουμε για την παρέμβασή σας αυτή. Και τώρα νίκ Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η πολλοί συνάδελφοι σε αυτή τη συζήτηση ε, έχουν ε, ομιλήσει και γενικά έχουμε αφιερώσει χρόνο. Εκ μέρους των Ευρωπαίων Συντηρητικών να πω ότι είμαστε υπέρ της απλούστευσης των κανόνων, όχι κατά αυτής. Θέλουμε η γραφειοκρατία να μειωθεί. Να υπογραμμίσω κάτι που παραγνωρίστηκε σε αυτή την συζήτηση και το ανέφερε ο όταν ε, μας παρουσίασε το θέμα. Ε, για, την υιοθέτηση όχι πλέον δεσμευτικών κανόνων μέσα από τη ε, διαδικασία της επιτροπολογίας. Αρίας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε να ευχαριστήσω το για όσα μας είπε που ήταν πολύ καλή δουλειά και να κάνω μερικά σχόλια. Ακούσαμε αρκετές απόψεις από όλους όσους πήραν το λόγο. Να πω και εγώ την δική μου άποψη πρώτα απ' όλα για την εναρμόνιση. Το είπα μερικές φορές, θα πρέπει να είναι μια οδηγία που να αφορά κυρίως ε, όχι μόνο τα κράτη που υπάρχουν ε, τα δικαιώματα και εκτιμένα του καταναλωτού, αλλά και όσα δεν υπάρχουν παρόμοια. Μια εναρμόνιση, μια κοινή, ένας κυλάχιστος κοινόμος παρανομαστής και σεβόμενοι και όσους ε, όσα κράτη δεν διαθέτουν, ας το πούμε έτσι, να Και γι' αυτό θα πρέπει ακριβώς ε, να δούμε πώς έχει η κατάσταση. Και ενημέρωση του καταναλωτήου επίσης, όπως αναφέρθηκε, είναι πολύ σημαντικό και ο καταναλωτής να μπορεί να ενημερώνεται κατάλληλα για τα δικαιώματά του τα ευρωπαϊκά και σε κάθε κρατός μέλος να προσπαθήσουν να ενημερώσουν τον καταναλωτή για το δικαιώματά του. Μια αναφορά επίσης σημαντική στο ηλεκτρονικό εμπόριο για το ηλεκτρονικό εμπόριο εδώ που είπαμε και για την Επιτροπή αυτά θα πρέπει να εξεταστούν. Το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν είναι το ίδιο όπως το παραδοσιακό εμπόριο. Στο τέλος βέβαια πωλείται ένα προϊόν. Είναι όμως κάτι διαφορετικό γιατί ο τρόπος διεξαγωγής εμπορίου είναι διαφορετικός. Και γι' αυτό ακριβώς αυτά θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα πλαίσια αυτής της οδηγίας, αλλά και με μια κάποια διαφοροποίηση, γιατί παραλαμβάνει κάτι διαφορετικό από ό,τι μέχρι σήμερα γνωρίσαμε. Αυτό θα πρέπει να εμφανιστεί ανάγλυφα και να το προσέξουμε περισσότερα. Δεν είναι αυτό για το ίντερνετ ε, παραξηγιακά κανενός ε, θα πρέπει να αναφερθεί και αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να προστατεύσουμε τα δικαιώματα του καταναλωτού στο ηλεκτρονικό εμπόριο ακριβώς, επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά. Θα πρέπει να προσέξουμε επίσης τις ε, διάφορες ε, απόψεις, πώς αντιμετωπίζει ο καθένας στη χώρα του τα πράγματα αυτή τη στιγμή της εναρμόνισης. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αυτό που είπα ότι είναι ένας ελάχιστος κοινοπαρομαστής έστω. Αλλά θα πρέπει να υπάρξει τουλάχιστον αυτά τα ελάχιστα να υπάρξει εναρμόνιση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ σημαντικό είναι ένας κατανοητής να μπορεί να ταξιδεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να γνωρίζει ε, και στην Ισπανία και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα τι δικαιώματα έχει από τη στιγμή που θα αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα και ε, ακόμα και όταν ε, μετατοπιστεί, ας το πούμε έτσι, γεωγραφικά. Αυτά ήθελα να πω σχετικά με τα μέχρι τώρα σχόλια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει και η Πρόεδρος. Ευχαριστούμε τον κύριο Αρίας και τώρα το λόγο έχει ο η κυρία Στάιλερ. Κυρία Στάιλερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους Κιώδης και τον εισηγητή. Νομίζω ότι δόθηκε πολύ τροφή για σκέψη μέσα από αυτές τις συζητήσεις. Καμιά φορά κάνουμε και κύκλους στη συζήτηση και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές ε, οπτικές γωνίες, είτε είναι πολιτιστικές είτε γλωστικές ε, Καμιά φορά όταν μιλάμε για το ηλεκτρονικό εμπόριο ξεχνάμε και αυτούς που δεν έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ και αυτοί πρέπει να προστατεύονται. Να τον αναγνωρίσουμε και αυτό. Υπάρχει και συζήτηση για τη μελέτη επιπτώσεων και ήθελα να μάθω αν έχει γίνει κάποια συζήτηση, αν έχει γίνει κάποια περαιτέρω αξιολόγηση επιπτώσεων, έτσι ώστε να δούμε ποια θα είναι τα ωφέλη και εναλλακτικέ λύσεις. Για την στοχευμένη εναρμόνιση νομίζω ότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από το γεγονό ότι οι τρέχουσες προτάσεις, ειδικά στα δική μου εκλογική περιφέρεια με τα, με τα δικαιώματα basic που έχουν, τα βασικά δικαιώματα, δηλαδή όπως το δικαίωμα απόρριψης. Αν ε, ακολουθήσουμε αυτή την οδό δεν θα έχουν αυτά τα δικαιώματα και αυτό τους ανησυχεί επίσης ε, η μείωση των υποχρεωτικών πληροφοριών που δίνονται στους καταναλωτές για τα προϊόντα τα χρηματοπιστωτικά, χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Πρέπει να διασφαλίσουμε την προστασία αυτών των ανθρώπων, αυτών των καταναλωτών. Χαίρομαι λοιπόν για αυτήν την συζήτηση. Χαίρομαι ε, που συζητούμε ε, για τα δικαιώματα των καταναλωτών και πρέπει να είναι συμπληρωματικά αυτά, συμπληρωματικές οι προσπάθειές μας. Ελπίζω Ε, ότι θα υπάρχει κάποια κίνηση γιατί σε όποια κατεύθυνση και να πάμε θα πρέπει κατά κύριο λόγο να έχουμε στο μυαλό μας την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Ευχαριστούμε. Ε, ε, ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ νομίζω ότι η συζήτηση σήμερα το πρωί ήταν ιδιαίτερα καρποφόρα. Άκουσα πάρα πολλές απόψεις, είχα ήδη ακούσει στην Επιτροπή, αλλά άκουσα σήμερα και τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Για πρώτη φορά φάνηκε κάτι πεντακάθαρα. Μας είπαν αρκετοί ότι αυτή η πρόταση δεν μπορεί να εφαρμοστεί με τη σημερινή μορφή. Χρειαζόμαστε σημαντικές αλλαγές της πρότασης. Κύριε ε, απευθύνομαι σε εσά. Η ερώτησή μου είναι πώς θα πετύχουμε βελτιώσεις για τον καταναλωτή. Καλό μήπως όμως θα ήταν από την αρχή να κάνουμε κάτι και για το εμπόριο μέσω ίντερνετ και έτσι έμεσα να ενισχύσουμε και σε άλλους τομείς τα δικαιώματα των καταναλωτών. Ίσως ε, όλα αυτά, όχι στα πλαίσια μιας πολύ μεγάλης οδηγίας, αλλά τουλάχιστον άμεσα στους κατανοτές και σε εταιρείε και στο διαμεθεριακό εμπόριο να απευθύνονται. Ε, ίσως θα ήταν και ένας καλός τρόπος αντιμετώπιση αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εσάς, σας ευχαριστώ πολύ. Κανέν, Με αρμοδιοσύνη για το θέμα αυτό. Κυρία Πίτικανεν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, λυπάμαι γιατί άργησα λιγάκι. Νομίζω ότι η θέση της ΕΚΟΝ συνάδει με αυτά που ακούσαμε σήμερα. Η βασική προσέγγιση είναι ότι ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παρέχει υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Αυτός είναι ο στόχος της οδηγίας, η εγγύηση υψηλού επίπεδου προστασίας και μία αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς έτσι ώστε να προωθηθεί η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο όλα αυτά τα θέματα να τα ευθυγραμμίσουμε, να τα συνδυάσουμε, γιατί αν είναι κατανοποιημένοι οι καταναλωτές θα είναι καλύτερη και ανταγωνιστικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσωπικά θεωρώ ότι χρειάζεται να προχωρήσουμε προσεκτικά, με προσεκτικά βήματα σε αυτό το θέμα της προστασίας των καταναλωτών. Η Κομισιόν θέλει πλήρη εναρμόνιση, αλλά μάλλον δεν θα μπορέσει να δουλέψει με αυτό το μοντέλο. Γιατί κανένα σκοπό δεν θα εξυπηρετήσει ούτε την υψηλότερη προστασία των καταναλωτών, ούτε μια πιο αποτελεσματική εσωτερική αγορά. Νομίζω ότι μάλλον προβλήματα θα δημιουργηθούν. ειδικότερα εκεί που υπάρχουν ε, συγκρουόμενες εθνικές νομοθεσίες. Έτσι λοιπόν υπάρχουν διάφοροι τομείς τελικά που μπαίνουν στο παιχνίδι. Για παράδειγμα, αν δούμε τι γίνεται με τα κινητά τηλέφωνα. Μπορεί κανείς να καταναλώνει όχι μόνο τηλεφωνικές υπηρεσίες, αλλά και μουσική μέσα από αυτά. Και αυτό πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας όταν υπογράφουμε συμβόλαια αυτού του είδους. Έχουμε νέες καινοτόμες χρηματοπιστωτικές ε, υπηρεσίες, ειδικότερα για τα υλικά αγαθά. Ε, όταν αυτό οδηγεί σε υλικά αγαθά, μάλλον θα πρέπει στο μέλλον να υπάρχουν ε, ξεχωριστοί κανόνες για τα χρηματοπιστωτικά. Για παράδειγμα, ένα μικρό δάνειο για ένα κινητό. Υπάρχουν νέοι καινοτόμοι τρόποι να αγοράσει κανείς μετοχές, αυτοκίνητα ή τη χρηματοδότηση της αγοράς αυτοκινήτων. Όλα αυτά ε, θα πρέπει να τα εξετάσουμε, να υπάρχουν λογικοί όροι στις συμβάσεις και να διασφαλίσουμε ότι όταν μιλάμε για νέα προϊόντα να κοιτάμε από πριν ποια τα προβλήματα και όχι μετά, αφού προκύψουν. Ε, τίθεται ένα υψηλό επίπεδο ντεμίνιμης από την οδηγία. Για τα μικρότερα, ας πούμε, δάνεια που διατίθεται με τους καινοτόμους αυτούς τρόπους μέσα από άλλους καινούριου ε, δρόμους ας πούμε. Να σας ευχαριστήσω για τα σχόλιά σας. Και να πω ότι θα σας στείλω τις πληροφορίες που έχουμε εδώ συλλέξει με βάση την εργασία μας επί της νομοδότησης. Πρέπει να προχωρήσουμε βήμα προς βήμα έτσι ώστε να δημιουργήσουμε υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και αυτό είναι και ο στόχος της νομοθεσίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εσάς. Η Επιτροπή έχει το λόγο. από το περιβάλλον της Επιτροπού Ρέντι. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι σήμερα υπάρχουν μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων εδώ. Το θέμα είναι ενδιαφέρον. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκφράσει ήδη το ενδιαφέρον του. Ευχαριστώ ιδιαίτερα λοιπόν και τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού αλλά και των Εθνικών Κοινοβουλίων για τη μέχρι τώρα συνεισφορά τους. Η συζήτηση είναι ενδιαφέρουσα, είναι ζωντανή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκοπός μας είναι να φτάσουμε σε ένα σύγχρονο τρόπο αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό και η Επίτροπος αποφάσισε να ακούσει και να συγκεντρώσει όλες τις απόψεις και τις ιδέες. Η Επιτροπή πρέπει να σας πω ότι εδώ και τέσσερις μήνες η Επιτροπή δεν λειτουργεί 100% πήρε περισσότερο χρόνο από ότι είχε αρχικά προβλεφθεί η όλη διαδικασία αλλά πραγματικά θέλω να σας καθησυχάσω. Θα ενισχύσουμε όλα τα κενά, θα προσπαθήσουμε μέσω στενής συνεργασίας μεταξύ Επιτροπής, Κοινοβουλίου και Συμβουλίου να δημιουργήσουμε μια καλύτερη πρόταση. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κύριο Σφάπ για τις προσπάθειές του, για το ότι όλα τα σημεία που αναφέρετε στην έκθεσή σας είναι εξαιρετικά σημαντικά σημεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Επίτροπος, αναρωτήθηκε πώς θα κάνει τους Ευρωπαίους καταναλωτές να νιώσουν άνετα με αυτή την πρόταση. Να νιώσουν οικία, οικειότητα. Εναρμόνιση. Εναρμόνιση για την εσωτερική αγορά. Τι άλλαξε από τη δεκαετία του 90 μέχρι σήμερα. Γνωρίζουμε τις παλιές οδηγίες με το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την προσπάθεια να δημιουργήσουμε μια συνεκτική οδηγία. Ακούγοντας όλους όσους πήραν το λόγο σήμερα, η απάντηση είναι σαφής. Αυτό που άλλαξε είναι το ίντερνετ, είναι το διαδίκτυο, είναι η δυνατότητα σήμερα να χρησιμοποιήσουμε νέους τρόπους και νέες τεχνολογίες. Άρα, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές, οι οποίοι βλέπουν κάτι σήμερα στο ίντερνετ και δεν μπορούν να το αποκτήσουν, γιατί, γιατί κάποιος, κάποια αριθμιστική αρχή τους λέει όχι, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Η νομοθεσία για τον Ευρωπαίο καταναλωτή, αν θέλετε με φυσικό τρόπο, θα πρέπει να οδηγήσει προς μία εναρμόνιση, πλήρη εναρμόνιση, στοχευμένη εναρμόνιση. Στην παρούσα πρόταση η πρόθεση ήταν να φτάσουμε σε μια στοχευμένη εναρμόνιση. Το θέμα όμως είναι να ε, αντιμετωπίσουμε όλες τις πτυχές και όλα τα επίπεδα αυτής της στοχευμένης εναρμόνισης. Σε πολλές χώρες κινδυνεύουμε να αποτύχουμε αν δεν αντιμετωπίσουμε τις πραγματικές ανάγκες των καταναλωτών. Και αυτό θέλει να αποφύγει η κυρία Ρέντινγκ. Αυτή είναι η γενική κατεύθυνση. Για τις λεπτομέρειες θα συζητήσουμε αργότερα. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Εδώ αλλάζουν οι πρόεδροι, όπως είδατε. Είμαι ο Μάικλ Χάρμπορ. Ζητώ συγγνώμη, είμαι ο πρόεδρος αυτής της Επιτροπής. Είμαι συντηρητικός μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα ήθελα για όλους όσους δεν με γνωρίζουν να σας χαιρετήσω. Σήμερα το πρωί στις 6 το πρωί ήμουν στη Φραγκφούρτη, στο αεροδρόμιο και πρέπει να σας πω ότι ήταν εξαιρετικά δύσκολο να φτάσω μέχρι εδώ. Ξέρω όμως ότι έχω πολύ καλούς αντιπροέδρους οι οποίοι έκαναν αυτό που έπρεπε στη θέση μου. Ξέρω επίσης ότι μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων πήραν ήδη το λόγο, ότι μίλησαν και οι Ευρωβουλευτές. Δεν ξέρω αν κάποιος θέλει να ξαναπάρει το λόγο, να απαντήσετε σε κάτι που ακούσατε, κάτι που σας ξάφνιασε. Ξέρω ότι μίλησε και ο εισηγητής, θα ξαναπάρει το λόγο. Ακούστηκε η έννοια της στοχευμένης εναρμόνισης. Το ερώτημα είναι, όταν έχουμε στόχους, ποιοι είναι οι στόχοι αυτοί, πώς ορίζονται στο περιεχόμενό τους και βεβαίως αυτό είναι πλέον πολιτικό θέμα. Με μεγάλη χαρά λοιπόν θα δώσω το λόγο σε όποιον από εσά θέλει να τον πάρει ή να τον ξαναπάρει. Αλλά ακριβώς επειδή έχουμε προσκεκλημένους από τα Εθνικά Κοινοβούλια, θα ήθελα καταρχήν να απευθυνθώ σε εσά. Δεν βλέπω τα ονόματά σας, δεν βλέπω τόσο μακριά, αλλά βλέπω ότι είστε από την Πολωνία. Ναι, είμαι από την Γερουσία της Πολωνίας και θα ήθελα πολύ σύντομα να αναφερθώ σε κάποια από τα σημεία που ακούστηκαν. Ανάλυση αντικτύπου πρέπει να γίνει σε τρεις τομείς. Πρώτον, στο νομικό, οικονομικό και κοινωνικό. Ακούστηκαν ε, πολλοί και διαφορετικοί τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος εδώ στην αίθουσα και πιστεύω ότι κάτι πολύ σημαντικό είναι η σταθερότητα των νομικών λύσεων που θα προτείνουμε με σκοπό να αποφευχθούν κενά, αδυναμίες και έλλειψη συνοχής που συνεχίζει να υπάρχει στις εθνικές νομοθεσίες. Δεύτερον, ο οικονομικός τομέας. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ο καταναλωτής, ο πολιτής, ο παραγωγός και οι σχέσεις μεταξύ αυτών των ε, διαφορετικών παραγόντων. Θα πρέπει αυτά να θεσμοθετηθούν. Τέλος, τα κοινωνικά, αν θέλετε, στοιχεία. Και εδώ δεν αναφέρομαι μόνο στο ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά σε οποιαδήποτε μεταφορά προϊόντων, όλες αυτές οι διαδικασίες θα πρέπει να εναρμονιστούν και τουλάχιστον να συμφωνήσουμε σε κοινού κανόνες. Η κοινωνική πτυχή όλων αυτών των αποφάσεων θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και να αναρωτηθούμε ποια είναι, αν θέλετε, η συνέπεια μιας πλήρους εναρμόνισης. Θέλουμε αυτήν την πλήρη εναρμόνιση. Για μένα η μεικτή, όπως θα την ονομάσω εναρμόνιση, είναι η ιδανική λύση. Νομίζω ότι ακούσατε ότι για πρώτη φορά οργανώθηκε μία συνδιάσκεψη μέσω βίντεο με την ε, συνεδρίαση για την προστασία του καθλό. Κυρία Καναμαλή, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Κυρία Καναμαλή, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιθυμούσα και πάλι το λόγο μετά από τις ανταλλαγές απόψεων αυτές που δείχνουν ότι αυτό που προδιαγράφεται τώρα μετά από την πρώτη συζήτηση τι είναι επιθυμούμε την πρόοδο χρειάζεται βέβαια ο απαραίτητος χρόνος θα πρέπει να ξεκινήσουμε από μια ελάχιστη εναρμόνιση από τα κεκτημένα είδη και σιγά σιγά να συμπληρώνουμε. Στη φάση αυτή να υποβάλω δύο ερωτήσεις και μία ερώτηση για τη μέθοδο. Πρώτο ερώτημα κύριε Επίτροπε, κύριε Συγητή. Λέτε αυτές τι καταχρητιστικές ρήτρες στα πρώτα λόγια που είπατε και ένα ενιαίο κατάλογο που αλλάζει μέσω της επιτροπολογίας αυτό όμως δεν είναι το κατάλληλο, δεν μπορεί να γίνει δεκτό. Μήπως ε, ευρωπαϊκοί κοινοί κατάλογοι που θα εμπλουτίζονται βαθμιαία από τους εθνικούς καταλόγους που εφαρμόζονται από όλα τα κράτη-μέλη συμπληρωματικά με όσα ήδη υπάρχουν. Ε, σε αυτό το σημείο νομίζω θα αποτελέσει πρόεδρο, πρόοδο και με ιδιαίτερη προσοχή άκουσα τους ε, διαφόρους που έλαβαν το λόγο, ε, Ρόιτοβα, την κυρία Ράπτη επίσης, ε, που αντιμετώπισαν το θέμα αυτό σχετικά με τις μελέτες εφικτού και είχαμε συγκροτηματικό πίνακα το Σεπτέμβριο του 2009 για τις συγκρίσεις μεταξύ κρατών μελών μετά από την πρώτη μου ανάγνωση είναι κάτι που δεν είναι επαρκές και επειδή ακούγονται διάφορα θέματα σήμερα μήπως καινούριε μελέτες ε, το τι ακριβώς γίνεται, τι σημαίνουν όλα αυτά για να δούμε για τη μέθοδο και το χρονοδιάγραμμα επίσης είναι σημαντικό στοιχείο και σημείο αν έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα που να αφορά μια μακρά χρονική περίοδο για την εφαρμογή του κειμένου θα ήταν κάτι το ιδιαίτερα θετικό και θα διευκόλυνε τις εργασίες μας. Κύριε Πρόεδρε σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Καραμαλή. Κάποιο άλλο μέλος Εθνικού Κοινοβουλίου θα ήθελε να πάρει το λόγο. Έχουμε τη δυνατότητα για έναν επιπλέον γύρο. Ναι, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δεν θα ήθελα εξ Γαλλίας να μονοπολίσουμε το λόγο εδώ, αλλά αποφελούμε μια και δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος ομιλητής. Εδώ αυτό το θέμα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Γαλλικό Κοινοβούλιο και σε άλλα κοινοβούλια δεσμευτική νομοθεσία είναι σβάρος η πραγματικότητα, το άκουσα σαν θέμα από όλου. Στην δική μου περίπτωση και αρκετοί Γάλλοι το πιστεύουν αυτό, ότι είναι το αντίθετο. Εάν δεν είναι δεσμευτική, τότε οι λιγότερο τίμιες επιχειρήσεις σε ευνοούνται απέναντι στις τίμιες επιχειρήσεις. Πάνω σε αυτό χρειάζεται να εργαστούμε, το συζητήσαμε ιδιαίτερα στη Γαλλία πριν από τέσσερα χρόνια για, την, για τον εύθερο ανταγωνισμό Χωρί τρέβλωση. Η στρέβλωση αυτή μπορεί να επέλθει μέσω νόθευσης των ρυθμίσεων και μάλιστα των ρυθμίσεων εκείνων που δεν γίνονται σεβαστές. Ωραία. Θέλει κάποιος άλλος να μιλήσει. Ανοίγω τον κατάλογο των ομιλητών για τα μέλη της Επιτροπής που θέλουν να συμβάλουμε νέες ιδέες και μετά θα δώσω την δυνατότητα στον κύριο ε, Σβάμπ να απαντήσει. Η κυρία Ρόιτοβα και η κυρία Γκέπχαρτ. Χωρίς μικρόφωνο. Μιλήτρια, δεν ακούγεται. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ φρέσκος φαίνεστε που ήρθατε από τη Σιγκαπούρη. Να χρησιμοποιήσω το χρόνο μας όμως και να καταθέσω άλλο ένα θέμα. Ο κύριος Φάπ το ανέφερε, αλλά ήθελα λίγο να παραμείνουμε. Σχετικά με τις μαύρες ή λίστες. Τεράστιο θέμα. Σας ζητώ λοιπόν να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Κάτι άλλο. Έχουμε την επιλογή επαναχώρησης από σύμβαση που ε, έχει ξεκάθαρες εγγυήσεις, ξεκάθαρους όρους. Για το διασυναρρογικό εμπόριο, ίσως δεν τον έφεραν οι συνάδελφοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια, αλλά συμφωνούμε σε αυτό. Στο επίπεδο εναρμόνισης έχουμε de minimis εναρμόνιση και θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε maximum εναρμόνιση. Αυτή είναι η πρόταση της Κομισιόν. Αυτή τη στιγμή θέλουμε να βρούμε μια συμβιβαστική λύση η οποία θα μας δώσει maximum εναρμόνιση σε σχέση με θέματα που δεν είναι αντιφατικά που δεν μειώνουν τα στάνταρ και τα όρια στα κράτη-μέλη και ταυτόχρονα να μην δημιουργήσουμε μία δίσκαμπτη και πολύπλοκη νέα νομοθεσία. Ξέρουμε ότι αυτό είναι καθήκον στη δική μας επιτροπή αλλά και καθήκον των επισκεπτών μας από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Πρέπει λοιπόν να δούμε πού είναι οι διαφορές, πού υπάρχουν παρεκκλήσεις. Θα ζητήσω για παράδειγμα στους Γερμανούς συναδέλφους, ε, η κυρία Γκέπχαρτ π.χ. να μας πει ποιες είναι οι διαφορές. Συνήθως έχουν υψηλότερα στάνταρ από τα ευρωπαϊκά. Φυσικά έχουμε λίγο διαφορετικές απόψεις και για την εγγύηση, την περίοδο εγγύησης. Αν έχετε μεγαλύτερη περίοδο εγγύησης, αυτό αντικατοπτρίζεται και στην τιμή των προϊόντων. Αν θέλετε, εγγύηση 3 με 5 χρόνια πληρώνετε παραπάνω. Αυτό είναι λογικό. Αλλά είναι και στρατηγική εταιριών που προσφέρουν ε, προϊόντα υψηλής ποιότητας. Μπορούν να ε, επιμικίνουν την ε, περίοδο της εγγύησης. Αυτό πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε, να το συζητήσουμε, να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών, ενημερωτικές εκστρατείες, έτσι ώστε οι καταναλωτές να γνωρίζουν πώς να διαβάζουν τις στρατηγικές των εταιριών. Αυτές οι στρατηγικές είναι καλές και για τους καταναλωτέ και για το διασυνοριακό εμπόριο. Και να θέσουμε και κάποια κοινά, ε, κάποιες κοινέ βάσεις, γιατί σε αυτό το τομέα θα βελτιωθούν τα στάνταρτα αν έχουμε κοινή βάση. Δίνω το λόγο στην κυρία Γκέπχαρτ, αλλά να πω ότι και η κυρία Ράπτη και η κυρία Κανέτη ζήτησαν το λόγο. Κυρία Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, μου δίνεται ευκαιρία να δώσω μία συμπληρωματική απάντηση. Κοιτάξτε, στην Γερμανία δεν είναι καλύτερη η κατάσταση σε σχέση με άλλα κράτη-μέλη για όλους τους τομείς που συζητούμε. Αυτό που μας απασχολεί εδώ να δούμε ποια είναι η κατάσταση στο κάθε κράτος μέλος ανάλογα με τον τομέα, το προϊόν ή την πτυχή που εξετάζουμε. Και αυτό θα δούμε σε πολλά παραδείγματα ότι διαφέρει. Είναι τελείως διαφορετική η κατάσταση από τον ένα τομέα στον άλλον. Ένα παράδειγμα, παραδείγματος χάρη, οι προθεσμίες για την επιστροφή. Η Επιτροπή προτείνει να υπάρξει πλήρης εναρμόνιση για κάποια προϊόντα, παραδείγματος. Να υπάρχει ε, προθεσμία δύο εβδομάδες ε, για κάποιες ε, συναλλαγές και αυτόματα να υπάρχει μια επέκταση αυτής της προθεσμίας για τρεις μήνες. Στη Γερμανία η προθεσμία αρχίζει να τρέχει από τη στιγμή όχι που υπεγράφει η σύμβαση, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει η αμφισβήτηση. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε άλλες χώρες όπως την ε, Τσεχία εάν παραδείγματο χάρη μετά από δύο εβδομάδες δεν υπάρχει η ε, παραλαβή του προϊόντος και από τη στιγμή που αρχίζει η διαδικασία αμφισβήτησης, αυτομάτως η διαδικασία επιμηκύνεται και η προθεσμία επεκτείνεται σε δύο ή τρεις μήνες. Αυτό λοιπόν που πρέπει να γίνει εδώ είναι η Επιτροπή να κάνει μια εκτίμηση αναπερίπτωση για το τι συμβαίνει στο κάθε τομέα, στα κράτη-μέλη, έτσι ώστε να αποφύγουμε τα κακά της πλήρους εναρμόνισης. Και πραγματικά αυτό πρέπει να γίνει μέχρι τον Οκτώβριο. Αλλιώς δεν θα υπάρξει καμία ανάλυση αντικτύπου, καμία σωστή εκτίμηση των επιπτώσεων. Και ακριβώς αυτό σήμερα προσάπτουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι δεν είναι σήμερα σε θέση να μας δώσει πληροφορίες και υπάρχει εντύπωση, μπορεί αυτό να είναι λάθος, αλλά υπάρχει εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά κάποιο τρόπο πρότεινε την πλήρη αναρμόνιση χωρίς προηγουμένως να εξετάσει ποιες είναι οι επιπτώσεις. Αυτό είναι το πρώτο σημείο που ήθελα να δείξω. Το δεύτερο το οποίο αναφέρατε, και γι' αυτό και ζήτησα το λόγο, οι επαφές με τους οργανισμούς προστασίας του καταναλωτή είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και εγώ θα ήθελα να σας δώσω κάποια στοιχεία για γερμανικούς οργανισμούς προστασίας του καταναλωτή να μπορέσετε να έρθετε σε επαφή γιατί μόνο έτσι οι πληροφορίες που διαθέτουμε μπορούν να επαληθευτούν και να εξακριβωθούν. Θα ήθελα και κάτι άλλο να πω, κάτι που ανέφερε ο κ. Γκομπέρ. Χρειαζόμαστε κανόνες Χρειαζόμαστε ρυθμίσεις. Όντω η προστασία του καταναλωτή πρέπει να βασίζεται σε κανόνες. Η ελάχιστη εναρμόνιση είναι κάτι που θα βασίζεται σε κανόνες. Δεν πρόκειται να το κάνουμε χωρίς κανόνες. Ζητούμε όμως ένα ελάχιστο επίπεδο κανόνων και προστασίας του καταναλωτή που να ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί και πέρα ο καθένα μπορεί να αυξήσει το επίπεδο προστασία του καταναλωτή. Θα πρέπει όμως να θεσπίσουμε το επίπεδο αυτό κάτω από το οποίο απαγορεύεται να πάμε. Επουδενή λόγο αυτό δεν σημαίνει ότι σε μια χώρα η κατάσταση θα επιδεινωθεί. Όχι. Κοιτάξτε άρθρο προς άρθρο πρέπει να προσέξουμε έτσι ώστε να μην μειωθούν τα δικαιώματα προστασίας του καταναλωτή σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπάρξει επιδείνωση της κατάστασης. Σας ευχαριστώ. Uh, uh. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Γκέπχαρτ, κυρία Κανιέτη και κατόπιν η κυρία Ράπτη. Με μεγάλη χαρά θα δώσω το λόγο και σε μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων, εάν θέλουν να ξαναπάρουν το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, να ξεκινήσω με ένα τεχνικό πρόβλημα. Γιατί είμαι πλήρως μέλος, πλήρες μέλος της Επιτροπής και πάλι έχω πρόβλημα και δεν μπορώ να μιλήσω στη μητρική μου. Και γι' αυτό αυτά που λέω ε, δεν είναι ξεκάθαρα και σαφή. Καμία γλώσσα δεν αντικαθιστά τη μητρική μας. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Ευχαριστώ όλα τα μέλη του Εθνικού, των Εθνικών Κοινοβουλίων που είναι εδώ, αλλά και ειδικότερα τον κύριο Σφάμπ για την ενέργεια που έδωσε και αφιέρωσε στην όλη προσπάθεια συζήτησης για το επίπεδο εναρμόνισης το οποίο αυτή τη στιγμή μπορούμε να συμφωνήσουμε κατά τη συζήτηση με τους εκπροσώπους των κρατών μελών και με τους συναδέλφους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο ότι δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε πλήρη εναρμόνιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Εγώ είμαι μεταξύ αυτών που λυπούνται, γιατί ακριβώς αυτή η πλήρης εναρμόνιση θα δώσει όλη τη δυναμικότητα που χρειάζεται η εσωτερική αγορά αυξάνοντας τη δυνατότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να ανοιχτούν σε νέες αγορές, σε νέα κράτη-μέλη. Έτσι μόνο θα μειωθεί ο κατακαιρματισμός της ενιαίας αγοράς. Αυτοί που βασικά αποφελούνται από την εσωτερική αγορά είναι οι καταναλωτές ακριβώς. Γι' αυτό κατανοώ και συμπονώ τους καταναλωτές και τις ε, ε, ενώσεις των καταναλωτών που εκφράζουν ανησυχίες. Τα κράτη-μέλη ως μέλη της εσωτερικής αγοράς ε, θα πρέπει να βρούμε τέτοιο τρόπο ώστε να ε, παράσχουν ε, καλύτερες υπηρεσίες, καλύτερη ποιότητα στους καταναλωτές και χαμηλότερες τιμές. Έτσι θα κάνουμε την εναρμόνιση. Πρέπει επίσης να έχουμε στο μυαλό μας ότι η μακροπρόθεσμα, η αναρμόνιση θα αυξήσει την γενική ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν πολλά υπέρ και κατά της πλήρους εναρμόνισης. Όταν εξετάζουμε τις διαφορές και τις ιστερικές ιδιαιτερότητες των δικαιωμάτων των καταναλωτών και των νομοθεσιών, ειδικότερα σε ιδιαίτερους τομείς ε, που αφορούν τα διάφορα κράτη-μέλη και τα 27 κράτη-μέλη για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις βλέπουμε ότι είναι περιορισμένες, ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να υποφεληθούν από τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά. Αν εμείς οι Ευρωπαίοι λοιπόν να παραμείνουμε κολλημένοι στο εγώ μας, στο εθνικό μας εγώ και δεν έχουμε μια ισχυρή θέληση να ενισχύσουμε την ενιαία αγορά, τότε σύντομα θα είμαστε αντιμέτωποι με τη δυσάρεστη κατάσταση του να είμαστε σε δεύτερη μοίρα στον παγκόσμιο ανταγωνισμό που δεν σταματά ποτέ. Και αυτό είναι το υψηλότερο τίμημα που θα πληρώσουν οι καταναλωτές μας εξαιτίας της έλλειψης πολιτικής θέλησης να ληφθεί η σωστή απόφαση τη σωστή στιγμή. Κατανοώ ότι οι διαφορές μεταξύ μας είναι πολλές. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να επιδιώξουμε την πλήρη εναρμόνιση. Κατανοώ ότι αυτό δεν είναι δυνατό να γίνει με μιας, με μία απόφαση. Α γίνει βήμα προς βήμα, αλλά ας προχωρήσουμε τέλος πάντων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Κανιέτη. Να πω ότι γνωρίζουμε το θέμα της έλλειψης λετωνικών και εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση ώστε να μπορείτε τελικά να χρησιμοποιήσετε και εσείς τη γλώσσα σας. Θα γράψω στο Γενικό Γραμματέα του Κοινοβουλίου σε σχέση με αυτό. Θα το λύσουμε. Κυρία Ράπτη. Καλώς ήρθατε κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Ε, δύο-τρία πραγματάκια, ε, έτσι για να κλείσουμε αυτή την κουβέντα που κάνουμε τώρα. Πρώτον, αισθάνομαι μία πρώτη ικανοποίηση που άκουσα τον εκπρόσωπο της Επιτροπής να μιλάει για στοχευμένη εναρμόνιση. Θεωρώ ότι είναι ένα θετικό βήμα. Όμως το είδαμε, το ακούσαμε στα λόγια μένει η πράξη, που είναι και το κυρίως ζητούμενο. Το δεύτερο ζήτημα είναι ε, τα δικαιώματα των καταναλωτών, αλλά και η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά, ώστε η εσωτερική αγορά να είναι ζωντανή, να είναι αποτελεσματική και να λειτουργεί. Έτσι λοιπόν α, σκέπτομαι και προτείνω ενδεχομένως ε, μία μελέτη ίσως θα μπορούσατε να σκεφτείτε, να αναθέσετε κύριε Σουάπ, για το κατά πόσον, για παράδειγμα, το κόστος από τη μείωση, την ενδεχόμενη μείωση του επίπεδου προστασίας σε ορισμένες χώρες, αντισταθμίζεται από τα ωφέλη στη διευκόλυνση του διασυνοριακού εμπορίου. Και το τελευταίο, είναι το εξής. Ε, δεδομένου ότι αυτού του είδους οι συνεδριάσεις όπως αυτή που κάνουμε σήμερα ε, φαίνεται να έχουν πάρα πολύ μεγάλη ε, επιτυχία και να συμβάλλουν στη δουλειά μας, μήπως θα έπρεπε να σκεφτούμε μία αντίστοιχη και ανάλογη ανταλλαγή απόψεων και με τις οργανώσεις των καταναλωτών. Ευχαριστώ. Um, Ευχαριστούμε πολύ. Κάποιος άλλος συνάδελφος από την Επιτροπή Ιστορικής Αγοράς που θέλει να λάβει το λόγο ή κάποιος από το Εθνικό Κοινοβούλιο. Όχι. Τότε και εγώ ως πρόεδρος να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία αφόσον έχουμε χρόνο και να κάνω και εγώ κάποιες παρατηρήσεις και μετά θα ζητήσω από τον κύριο Σφάπ να συνοψίσει. Δεν ξέρω αν ο κύριος Πρόγκ θέλει να δευτερολογήσει. Ίσως και αυτός θέλει να μας πει κάποια πράγματα. Πριν δώσω τον τελευταίο λόγο στον κύριο Σφάμπ. Από όσα άκουσα ως τώρα και έχοντας δει και τις αξιόλογες εκθέσεις από τις διάφορες επιτροπές σας, που είναι πολύ ενδιαφέρουσες, είναι θέμα της μελλοντική μας συνεργασίας ότι σε κάποιες περιπτώσεις ναι μεν ε, προχωρούμε άμεσα αλλά θα πρέπει να υπάρχει ε, και αμοιβαιότητα να στέλνει και η Επιτροπή σας εμάς τις ε, εκθέσεις και το αντίθετο για να μπορούν τα μέλη να έχουν χωνέψει τα βασικά σημεία που έχετε θίξει πριν συζητήσουν δόθηκε μια ευκαιρία για ε, μία συνάντηση με την Επιτροπή για την Προστασία των Καταναλωτών στο Εθνικό Κοινοβούλιο της Γαλλίας. Ήταν πολύ επιτυχημένη αυτή η συνάντηση. Έγινε με βιντεο conferencing, έγινε και μεγάλη ανταλλαγή πληροφοριών. Υπάρχουν πολλά πράγματα που θέλουμε να αμοιβαία να συζητήσουμε. Μέσα στα πλαίσια της, ε, της δίκης της υπάρχει και αυτή η διαρθρωμένη διαβούλευση με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Αυτή η Επιτροπή κατά κάποιο τρόπο το προέβλεψε αυτό και ήδη, όπως θα έλεγαν και οι συγητές, έχουμε τη δεύτερη ανταλλαγή απόψεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια σε αυτό το σημαντικό θέμα. Τον περασμένο μήνα έγινε το και για την οδηγία με τις καθυστερημένες πληρωμές. Και σχεδιάζουμε και άλλες δύο ανταλλαγές απόψεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια, καθώς προχωρεί η νομοθεσία, γιατί κομμάτι της ευθύνης στην Επιτροπή μας είναι να αναθεωρήσουμε κάποια από τα πιο κρίσιμα ε, νομοθετικά εργαλεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον τομέα της ε, εσωτερικής αγοράς. Και όσον αφορά <clears throat> την εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας, πιστεύω ότι το επόμενο θέμα τον Οκτώβριο θα είναι η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Και βεβαίως μια σειρά προτάσεων υπάρχει. Θα πρέπει να εξετάσουμε και τις ε, επερχόμενες εφαρμοστικές διατάξεις, αλλά νομίζω ότι και εδώ η συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια είναι εξαιρετικά σημαντική. Τι άλλες προοπτικές έχουμε. Και εδώ μιλάω για την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Πρέπει να σκεφτούμε και εδώ η δέσμευση των Εθνικών Κοινοβουλίων είναι πολύ σημαντική είναι το θέμα της εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών είναι σημείο κλειδί σε όλη αυτή τη διαδικασία και σε όλο αυτό το εγχείρημα. Πρέπει η νομοθεσία να ενσωματώσει αυτή την αρχή της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, να την ενδυναμώσει. Πρέπει να βελτιώσουμε την κατάσταση. Γιατί κάτι το οποίο παρατηρούμε τον τελευταίο καιρό, όσον αφορά παραδείγματο χάρη την οδηγία για τις παράνομες εμπορικές πρακτικές και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που απασχόλησε όλες τις χώρες είναι ότι πραγματικά και ενώ δεν εφαρμόζονται οι διάφορες διατάξεις όπως πρέπει και ακριβώς επειδή δεν καταφέραμε να φτάσουμε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο εναρμόνισης θα πρέπει να δούμε εάν ναι ή όχι υπάρχουν προϋπάρχουσες διατάξεις. Εάν ναι ή όχι, παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οργανώσεις προστασίας των καταναλωτών έχουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο δράσης και προστασίας. Η εμπιστοσύνη λοιπόν των καταναλωτών είναι πολύ σημαντική και θα πρέπει να διακατέχει όλο το πνεύμα αυτής της οδηγίας. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι η διαδικασία για την καταναλωτική πίστη, η οδηγία για την καταναλωτική πίστη και η προσπάθεια εναρμόνισης, μεγάλης εναρμόνισης, κάτι που όπως ξέρετε απερίφθη από το Κοινοβούλιο. Ζητάμε και εδώ στοχευμένη δράση και ιδιαίτερα στον τομέα αυτό όπου χρειάζονται οι καταναλωτές σημαντική προστασία. Υπάρχουν όμως μεγάλες αλλαγές, μεγάλες διακυμάνσεις από τη μία χώρα στην άλλη και η κατάσταση εξελίσσεται ακόμα. Εργαζόμαστε λοιπόν από κοινού και επεξεργαζόμαστε δύο διαφορετικούς τομείς και κοιτάμε την αναρμόνιση και στα δύο αυτά θέματα. Είναι πολύ σημαντικό ακούγοντάς σας σήμερα Ξέρω ότι πολλοί συμφωνούν με αυτά που ακούστηκαν εδώ. Η απώλεια, η υποχώρηση αν θέλετε όσον αφορά κάποια δικαιώματα που υπάρχουν στις χώρες είναι κάτι που προκαλεί φόβο. Σήμερα και επανέρχομαι εδώ σε αυτό που είπε ο κύριος Πρόν και η Επιτροπή έχει συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα και ενδεχομένως θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια δομή η οποία να λαμβάνει υπόψη της τα υπάρχοντα δικαιώματα, το υπάρχον επίπεδο προστασίας και να μην εμποδίσει όλους αυτούς οι οποίοι θέλουν να ενσωματωθούν στην αγορά και ιδιαίτερα εδώ μας ενδιαφέρουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 27 διαφορετικά νομικά συστήματα και νομοθεσίες. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε περαιτέρω προβλήματα και εμπόδια. Αυτά λοιπόν είναι τα θέματα που καλούμαστε να συζητήσουμε σήμερα. Και κατά την άποψή μου, ένα δύσκολο θέμα θα είναι ότι επεξεργαζόμαστε το θέμα αυτό χωρίς συγκεκριμένη στρατηγική πλαισίωσης. Μιλάμε για εναρμόνιση. Μιλάμε για εναρμόνιση της προστασίας των καταναλωτών. Πού πάμε. Ξέρετε ότι σήμερα έχουμε μπροστά μας ένα παζλ. Και κύριε Πρόγκ, αυτά που ακούστηκαν εδώ, και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα, πρέπει να μεταφερθούν στο γραφείο της Επιτρόπου. Το θέμα της αγοράς online. Κάτι το οποίο θέλουν οι καταναλωτές να το αντιμετωπίσουμε, να το επεξεργαστούμε με ρεαλιστικές λύσεις. Σήμερα υπάρχει ασάφεια προσφορά προϊόντων, υπηρεσιών με διαφορετικά νομικά συστήματα, αναφορετικές νομοθεσίες. Η έλλειψη εναρμονισμένου πλαισίου σήμερα δημιουργεί περισσότερα ερωτηματικά και προβλήματα με τις νέες τεχνολογίες. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε στρατηγικά το θέμα, να επεξεργαστούμε την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών, να συμφωνήσουμε που όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση και από εκεί και πέρα να δούμε αν για τις, το εμπόριο online μπορεί να υπάρξει ένα ειδικό καθεστώς. Με ερωτηματικό το λέω αυτό. Για να υπάρξει πραγματική προστασία των καταναλωτών. είναι πολύ πιο δύσκολο για έναν καταναλωτή να κάνει επιλογές, να νιώσει εμπιστοσύνη, να νιώσει ότι μπορεί να επιστρέψει παραδείγματο χάρη ένα προϊόν το οποίο αγόρασε online από την άμεση εμπορική επαφή που έχει ο καταναλωτής με τον πολιτή στο παραδοσιακό εμπόριο. Πιστεύω λοιπόν ότι τα ψηφιακά προϊόντα είναι και αυτό ένα θέμα που ανέφεραν πολλοί σήμερα το πρωί, αλλά και η εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας. Και εδώ θα ξανά αναφερθώ στην οδηγία για την καταναλωτική πίστη. Ξέρω ότι πολλοί έχετε εργαστεί για το θέμα αυτό, αλλά και στο θέμα της καταναλωτικής πίστης υπάρχουν πολλά προβλήματα. Δάνεια, παραδείγματος χάριν, που προτείνονται και αναλαμβάνονται με ηλεκτρονικό τρόπο. Για όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε κοιτώντας και μη ε, ξεχνώντας τους στρατηγικούς στόχους. Ξέρω ότι η νέα πρόταση Επιτροπής θα μας ε, βοηθήσει, αλλά Υποψιάζομαι ότι πολλοί στο Συμβούλιο θα συμφωνήσουν με τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ελπίζω αυτά που είπα να μην είναι διαφορετικά από τα συμπεράσματα στο οποία φτάσατε πριν ξεκινήσω εγώ την Προεδρία. Θα ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Σφάμπ. Ο κύριος Πόντσιλος νομίζω θέλει να πάρει το λόγο και σας ε, τον δίνω αμέσως. Ίσως και η Επιτροπή θέλει να ξαναπάρει το λόγο πριν τελικά τον δώσουμε στον Ανδρέα Σφάμπ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αισθάνομαι ως θύμα. Είμαι ένας καταναλωτής ε, που έπεσε θύμα αργοπορίας μιας πτήσης. Γι' αυτό έφτασα αργά και ζητώ συγγνώμη. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μιλάμε για την οδηγία των καταναλωτών. Το θέμα είναι ποιος είναι ο γενικός στόχος αυτής της οδηγίας είναι η ικανοποίηση των καταναλωτών. Έτσι πρέπει να το εξετάσουμε. Εγγυόμαστε αυτή την ικανοποίηση ή όχι. Εάν αποφασίσουμε να εναρμονίσουμε και να συγχωνεύσουμε τέσσερις ε, οδηγίες σε μία θα αυξήσουμε την ικανοποίηση και ασφάλεια των καταναλωτών στην αγορά. Γνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει διάφορες πρωτοβουλίες και ίσως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να τις εξετάσει πιο στενά. Ίσως να αξίζει τον κόπο να εξετάσουμε τα έτοιμα το έτοιμο κείμενο της νέας οδηγίας και να το αναλύσουμε από την άποψη των πιο κοινών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στα κράτη-μέλη. Δεν εννοώ ότι ο καθένας μας θα πρέπει να είναι πλήρως ικανοποιημένος από κάθε ρήτρα σε αυτό το έγγραφο, αλλά ε, αν μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας τις ανησυχίες, τα παράπονα των καταναλωτών στα διάφορα κράτη-μέλη, θα μπορούμε να αξιολογήσουμε αν τελικά αυτή η οδηγία θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής τους. Κάτι άλλο εξίσου σημαντικό είναι ότι πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε ποιοι είναι οι τομείς που καλύπτονται από τα δικαιώματα των καταναλωτών. Με άλλα λόγια, πού υπάρχουν οι περισσότερες αδυναμίες. Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες είναι κάτι που θα πρέπει να ληφθεί περισσότερο υπόψη στην οδηγία αυτή μιλώ εκ μέρους μίας χώρας όπου το 90% ε, των ε, τραπεζών έχουν ιδιωτικοποιηθεί αφού τα αφού πριν είχαν κρατικοποιηθεί. Άρα είναι σημαντικό οι καταναλωτές να έχουν ίσα δικαιώματα. Όταν πηγαίνει κανείς στην τράπεζα να ανοίξει λογαριασμό, να πάρει ένα δάνειο, συνήθως παίρνει έναν κατάλογο πραγμάτων που πρέπει πρώτα να κάνουν και μετά άλλον έναν κατάλογο με χρεώσεις ε, που πρέπει να πληρώσουν. Νομίζω λοιπόν ότι οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες πρέπει να αντιμετωπιστούν από την οδηγία γιατί αποτελούν ζωτικό κομμάτι της καθημερινής μας ζωής σήμερα. Ένα άλλο θέμα. Η κατασκευή νέων σπιτιών, ε, βιομερισμάτων, οι μεταφορές, όπως σας είπα, σήμερα έπεσα θύμα. Ε, γιατί ε, καθυστέρησα να φτάσω σε αυτή την επιτροπή. Και κανείς δεν μου είπε τίποτα, ούτε εμένα ούτε στους άλλους, ούτε σε μένα ούτε στους άλλους επιβάτες ε, σχετικά με τη βλάβη που είχε το αεροπλάνο. Καμία εξήγηση δεν μας δόθηκε. Νομίζω λοιπόν ότι αν πρέπει να επεκτείνουμε την οδηγία και το πεδίο εφαρμογή τη, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τέτοια πράγματα όπω είναι οι τραπεζικέ υπηρεσίε και οι μεταφορέ. Για τι μεταφορέ και πάλι. Για παράδειγμα, μπορούμε να αγοράσουμε ένα πριν από την υπηρεσία που θα μας παρασχεθεί. Το εμπόριο, άλλη σημαντικός ε, κλάδος. Σε κάποιες χώρες της Ευρώπης δεν ε, επιστρέφονται τα χρήματα ε, αν επιστρέψει ένα προϊόν. Αν εξετάσουμε το τι γίνεται στην Πολωνία και τι γίνεται στην οδηγία, κάνουμε, είναι ένα βήμα πίσω. Ως τώρα, ε, εμείς μπορούμε να επιλέξουμε ε, ως ε, πελάτες πώς θα γίνει η επιστροφή ε, του προϊόντος και αν θα πάρουμε επιστροφή χρημάτων ή άλλο προϊόν. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα κατάλογο με τα ελάχιστα στα οποία συμφωνούν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν μιλάμε για εναρμόνιση. Εάν ένα κράτος μέλος έχει επιτύχει κάποια πράγματα στο τομέα των δικαιωμάτων των καταναλωτών θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Η μεικτή λοιπόν εναρμόνιση είναι ό,τι καλύτερο και για την Πολωνία και για τα άλλη κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ε, εγώ άργησα γιατί υπήρχε θέμα στις ε, σχέσεις, ε, της βιομηχανικές και όχι σε αεροπλάνο. Να πω ότι γενικά εδώ έχουμε δουλέψει πολύ για τα δικαιώματα των επιβατών. Είχατε δικαίωμα για πληροφόρηση και σε αυτό το θέμα έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο νομίζω. Οι συνάδελφοι από την Επιτροπή Μεταφορών επίσης εξετάζουν ε, το πώς θα βελτιώσουν τα δικαιώματα των ε, επιβατών των αεροπορικών εταιριών. Ωραία. Ο κύριος Πρόγκ θέλει να κάνει ένα σχόλιο νομίζω. Ε, τελευταία ευκαιρία να μιλήσετε. Κύριε Πρόγκ, έχετε το λόγο. Και μετά ε, ο Αντρέας Σβάμπ θα κάνει μία συνολική σύνοψη. Ο κύριος Πρόγκ, λοιπόν, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι πρέπει να κατανοήσουμε ότι έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια ήδη στο θέμα της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, της προστασίας. Οι αλλαγές πρέπει να γίνουν με μεγάλη προσοχή. Πίτροπος θέλει να κρατήσει στο επίκεντρο και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών αλλά και την εσωτερική αγορά εν μέσω της κρίσης που γνωρίζουμε σήμερα. Όλοι βεβαίως θέλουμε στην Επιτροπή να συνεχίσουμε τη συνεργασία με την δική σας Επιτροπή για να βρεθούν λύσεις δεν είναι αδύνατο να βρεθούν αυτές οι λύσεις. Παρ' όλα αυτά θεωρούμε ότι ήδη έχει γίνει πολλή προσπάθεια και έχει καταναλωθεί πολλή χρόνος και ενέργεια. Θα συνεχίσουμε την σκληρή μας εργασία, λέει ο Πρόεδρος. Μπορείτε να συνοψίσετε, κύριε Σφάπ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πίστευα πραγματικά ότι αυτή η ανταλλαγή απόψεων θα μας επέτρεπε να συζητήσουμε κάποια από τα σημεία. Θα προσπαθήσω λοιπόν να συνοψίσω. Πολλά θέματα τα οποία θεωρούνται λεπτομεριακά δεν τα συζητήσαμε σήμερα καθόλου. Πολλά από αυτά δεν τα συζητήσαμε καθόλου. Και για όλα αυτά τα θέματα χρειάζονται λύσεις. Σας ευχαριστώ για τα θέματα που θίξατε, αλλά επαναλαμβάνω υπάρχουν πολλά από αυτά τα οποία και ο Σκιώδης εισηγητής και εγώ αλλά και μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων θεωρούν ενδιαφέροντα, σημαντικά και τα οποία χρήζουν λύσεις. Βεβαίως, αν αρχίζει μια συζήτηση, ποτέ δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει. Πολλές φορές λοιπόν Ακούσαμε το επιχείρημα της πλήρους εναρμόνισης. Όχι, αυτή δεν την επιθυμούμε. Το θέμα είναι να τεθούν οι στόχοι, οι όσον αφορά αυτή την εναρμόνιση. Οι τομεί δηλαδή και το επίπεδο της επιθυμητής εναρμόνισης. Ο Μάικλ Χάρμπορ είπε ότι φυσικά χρειαζόμαστε στρατηγική. Σήμερα δεν υπάρχει ευρωπαϊκή, ε, αν θέλετε, αίτηση αίτημα ευρωπαϊκό για εναρμόνιση. Αυτό δεν είναι κάτι το ε, αυτόματο και την ίδια ώρα. Όταν ξεκινάμε με διαδικασία εναρμόνισης υπάρχουν δυσκολίες. Θα τα αναφέρω τα προβλήματα αυτά. Από την άλλη μεριά θα πρέπει από κοινού τις εθνικές αρχές να προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες αυτές και να βρούμε λύσεις. Αλλιώς τα προβλήματα θα παραμείνουν και οι λύσεις που θα βρεθούν δεν είναι αυτές που πρέπει σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Τα προβλήματα πρέπει να επιληθούν από κοινού μεταξύ παραδείγματο χάρη των εθνικών αρχών όταν δεν είναι αρμόδιο το ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό μπορεί να μην αρέσει πάντα στα κράτη-μέλη. Όμως, εκεί που το ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να είναι το καλύτερο, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών, ο τίτλος της οδηγίας είναι «Δικαιώματα των καταναλωτών». Και τα δικαιώματα αυτά θα πρέπει να υποστηριχτούν και να προστατευτούν στο υψηλότερο επίπεδο. Πρέπει να πετύχουμε εκεί που αυτό είναι δυνατόν ένα πολύ υψηλό επίπεδο προστασίας. Και δεν το λέω αυτό με αφέλεια. Το λέω γιατί πραγματικά αυτό περιμένει ο Ευρωπαίος καταναλωτής. Και εδώ έχουμε τη δυνατότητα στους τομείς αυτούς που θα επιλέξουμε να φτάσουμε σε πραγματική αναρμόνιση. Αυτό βεβαίως αναπερίπτωση και εξετάζοντας όλους αυτούς τους τομείς. Η κυρία Ράπτη πολύ σωστά είπε ότι αυτό πρέπει να γίνει συστατιακά. Αύριο ξέρω ότι θα υπάρξει η απόφαση των συντονιστών και θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η μελέτη και η κατεύθυνση που θα ακολουθήσουμε. Αυτό πρέπει να γίνει, επαναλαμβάνω, σταδιακά, κομμάτι-κομμάτι, τμήμα προς τμήμα και εδώ χρειαζόμαστε τη συνδρομή της Επιτροπής έτσι ώστε να δούμε ποια είναι η κατάσταση στον κάθε τομέα, στο κάθε κράτος μέλος και να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις. Για τις επόμενες διαπραγματεύσεις και συνομιλίες θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μιλάμε για την πρόταση της Επιτροπής έτσι όπως έχει υποβληθεί. Και αυτό δεν χρειάζεται να το επαναλαμβάνω. Σας υπόσχομαι ότι η νέα πρόταση θα υποβληθεί από μένα με τον σκιώδη εισηγητή. Θα ενσωματώσω όλα τα σημεία τα οποία συζητήσαμε εδώ μετά από εξέταση και αφού εξετάσουμε αν μπορούν να ενσωματωθούν στην ε, πρόταση ή όχι. Κυρία Τάκ, εγώ δεν καταλαβαίνω την ερμηνεία που δίνεται στο άρθρο 95 της συνθήκης. Πρόκειται για μία αποστολή, για μία εντολή η οποία σαφώς και δίνεται από τη συνθήκη της Λισαβόνας, κατά την άποψή μου, για την επίλυση προβλημάτων των Ευρωπαίων καταναλωτών. Αυτό βεβαίως κάνοντας ένα σαφή διαχωρισμό του τι είναι αρμοδιότητα του εθνικού και τι είναι αρμοδιότητα του ευρωπαϊκού επίπεδου. Δεν καθορίζονται όμως απλώς οι αρμοδιότητες ανά επίπεδο. Γιατί εδώ σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να απομακρυνθούν τα κράτη-μέλη από την οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ε, πρωτοβουλία. Είναι απαραίτητη η συνεργασία και η ανταλλαγή απόψεων. Γι' αυτό και θέλουμε να ενδυναμώσουμε στο μέλλον τις επαφές μαζί σας η ελάχιστη εναρμόνιση. Η ελάχιστη εναρμόνιση σαφώς και είναι καλύτερη από το τίποτα. Αλλά αυτή η ελάχιστη εναρμόνιση που υπάρχει σήμερα πρέπει σαφώς να βελτιωθεί και να επεκταθεί. Βεβαίως έχουμε μπει σε λεπτομέρειες. Το ερώτημα καταρχήν είναι ποιοι είναι οι τομείς που πρέπει να εναρμονίσουν και πριν όχι. Πρέπει να συζητήσουμε την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Η Ρωσάντα έκανε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση αν πρέπει παραδείγματο χάρη να ξεχωρίσουμε κάποιους τομείς τους οποίους να υπάρχει εναρμόνιση και κάποιους μέσω οδηγίας και κάποιους άλλους μέσω κανονισμού η ελάχιστη εναρμόνιση ουσιαστικά θέτει το κατώτερο όριο πάνω από το οποίο καλούνται τα κράτη-μέλη να διατηρήσουν το επίπεδο της προστασίας τους. Προς τα πάνω δεν υπάρχει όριο. Και αυτό που είναι σημαντικό είναι από εκεί και πέρα να υπάρχει παρακολούθηση και έλεγχος για το πώς αυτό το ελάχιστο επίπεδο τηρείται. Περισσότερη διαφάνεια λοιπόν, καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών, των Ευρωπαίων πολιτών για τα δικαιώματά τους έτσι ώστε να υπάρξει δυνατότητα προσφυγής, ελέγχου και επαφή. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν πρέπει να ξεχνάμε και το θέμα του οικονομικού κόστους. Βλέπουμε ότι εδώ οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι παρούσες στις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, έχουν δυνατότητες που οι μικρομεσαίες σήμερα δεν έχουν. Πρέπει όμως να δούμε και τις δυνατότητες που προτείνουμε σήμερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έτσι ώστε να προσαρμοστούν σε αυτά τα νέα δεδομένα της αγοράς. Ελάχιστη λοιπόν εναρμόνιση για αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που μέχρι τώρα δεν έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Τώρα, όσον αφορά κάποια κράτη-μέλη που παραμένουν στην εθνική τους παράδοση, η αναποτελεσματικότητα, να το πούμε έτσι. Αυτές οι παραδόσεις υπάρχουν, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν προσπαθούμε να τις ταρακουνήσουμε ή να τις ξεπεράσουμε. Και κάθε φορά πρέπει να αποδείξουμε τι είναι η πιο αποτελεσματική προστασία του καταναλωτή. Ποιο είναι το ευρωπαϊκό επίπεδο, αν είναι αποτελεσματικό και αν το εθνικό επίπεδο είναι λιγότερο αποτελεσματικό. Κάθε φορά λοιπόν θα πρέπει να γίνεται μια αναπερίπτωση εξέταση. Υπάρχουν όμως και θέματα και δυσκολίες και προβλήματα που δεν τα έχουμε συζητήσει, όπως παραδείγματος χάρη οι οδηγίες Ρώμη 1 και Βρυξέλλες 1. Θέλουμε μια εσωτερική αγορά η οποία να αυξάνει τις δυνατότητες να ξεπεραστούν τα εμπόδια και τα σύνορα. Και είχα πολύ ενδιαφέρουσες συνομιλίες με εκπροσώπους μικρών κρατών μελών, οι οποίοι έχουν την άποψη ότι παραδείγματος χάρη η δυνατότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σαφώς και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη με ένα διαφορετικό τρόπο σήμερα στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Η πρόταση την οποία θα πρέπει να προετοιμάσουμε θα πρέπει να υποστηριχθεί από την πλειοψηφία των πολιτικών ομάδων, από τα 27 κράτη-μέλη με 27 διαφορετικά νομικά συστήματα. Το θέμα της νομικής βάσης επίσης θα πρέπει να συζητηθεί. Ελπίζω η Επιτροπή να άκουσε πολύ προσεκτικά όλες τις απόψεις και να είναι στη διάθεση όλων των μελών της Επιτροπής μας. Και γνωρίζω ότι κυρία Γκέμπχαρτ σε κάποια σημεία μπορεί εσείς να έχετε δίκιο, σε κάποια άλλα ίσως να έχω εγώ. Ξέρετε πολύ καλά ότι η υπόθεση eBay μας έδειξε ότι η προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών οδηγεί πολλές φορές και σε αρνητικές συνέπειες. Το θέμα της προθεσμίας, ναι. Όντως πρέπει κατά την άποψή μου να υπάρξει εναρμόνιση. Κυρία Τάκ, είπατε ότι έχουμε τεχνικά εμπόδια. Μπορεί όμως το πρόβλημα να είναι και πολιτικό. Η πληθώρα των διαφορετικών ρυθμίσεων όντως δημιουργεί σήμερα πρόβλημα. Κυρία Καραμαλή, έχετε δίκιο όταν μιλάτε για την κρίζα μαύρη λίστα με τις επιτροπολογίες. Το θέμα όμως είναι ότι αυτές οι ρήτρε υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όπως είπε και ο κύριος Γκομπέρ, αυτοί οι οποίοι τηρούν τις ρυθμίσεις θα πρέπει να τη στηρούν όχι μόνο στη χώρα τους, αλλά σε όλη την Ευρώπη. Αυτές οι ρήτρε θα πρέπει σαφώς και να είναι εναρμονισμένες προς όφελος της διαφάνειας και της προστασίας των καταναλωτών. Σε μια παραδοσιακή εμπορική συναλλαγή υπάρχουν συγκεκριμένα δικαιώματα και ευθύνες των πολιτών και των αγοραστών. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η μαύρη λίστα συμπεριλαμβάνει μια παρόμοια ε, σειρά ε, ρυθμίσεων και ρητρών για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Χρειάζεται, χρειάζεται βεβαίως η δυνατότητα περισσότερης ευελιξίας έτσι ώστε να μπορούν να βρεθούν λύσεις και γι' αυτό και αναφέραμε και στο κεφάλαιο 5 όπου αναφέρονται τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις για όλες αυτές τις εμπορικές συναλλαγές που ξεπερνούν τα σύνορα έτσι ώστε να υπάρξει ένα εναρμονισμένο πεδίο στην Ευρώπη με ευελιξία και με τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε σημερινά προβλήματα. Τελειώνοντας κυρίες και κύριοι θέλω να σας πω ότι δικό μας καθήκον είναι να αντιμετωπίσουμε την πολυμορφία στην Ευρώπη, την πολυμορφία, την πολιτική, την τεχνική που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Ευρωπαίοι καταναλωτές. Ελπίζω η πρόταση που θα υποβάλουμε να συμπεριλαμβάνει όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν σήμερα. Είμαι αισιόδοξο. Θεωρώ ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η σημερινή συζήτηση. Θα σε ευχαριστώ πολύ και πιστεύω ότι σκοπό μα είναι και η εσωτερική αγορά αλλά και η προστασία των καταναλωτών, η οποία θα πρέπει να βελτιωθεί. Ευχαριστούμε πολύ, Αντρέα. Νομίζω ότι κάπου εδώ τελειώνουν οι σημερινέ μα εργασίε. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά όλοι τα μέλη του Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων και τις ομάδες υποστήριξη που ήρθαν εδώ σήμερα μαζί τους. Είστε πάντοτε πρόσδεκτοι για συμμετοχή στις μελλοντικέ ε, συνεδριάσεις μας. Θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε το πώς προχωράει η δουλειά μας. στην έκθεση του κυρίου Σφάμπ. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Πριν κηρύξω το πέρας της συνεδρίασης, να σας θυμίσω, να θυμίσω στα μέλη της Επιτροπής ότι το απόγευμα έχουμε πολλές πολύπλοκες ψηφοφορίες. Να φέρετε λοιπόν τις κάρτες σας μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ και ε, θα τα ξαναπούμε.